Morning, ladies and gentlemen. It's uh, και πέντε πήγε, λέει ο πρόεδρο. Ήδη, ήδη, ήδη αργήσαμε, οπότε ε, ε, θα ήθελα τώρα να αρχίσουμε τη συνεδρίαση με την έγκριση τη μεσαία διατάξεω. Ωραία, πριν όμω ε, την εγκρίνουμε, θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι σήμερα θα έχουμε και ένα δεύτερο τριμερή διάλογο για τις Προτιμήσει τι εμπορικέ σχέση με το Πακιστάν και αν προκύψει μια λύση ε, παρακαλώ να το κοιτάξουμε αύριο, να το βάλουμε στη διάταξη για την ψήφιση και τι ψηφορίε αύριο. Το 5 παρουσίαση Τον, ε, το, το 5 θα αναλυθεί τέλο πάντων που είναι η παρουσίαση των υπηρεσιών των μέσων ενημέρωση. Εντάξει με τα πρακτικά. Είστε όλοι ικανοποιημένοι. Τρία. Ανακοινώσει του Πρόεδρου. Θα ήθελα να σα ενημερώσω ότι μεταδίδεται μέσω του Ιντερνετ η συνεδρίαση και υπάρχει και κάτι άλλο. Ότι θα πρέπει να προσέχετε να πατάτε το κουμπάκι όταν θέλετε να μιλήσετε. Φαίνεται αυτονόητο, ναι, άλλο δεν είναι. Επίσης, έχετε λάβει τα σχετικά έγγραφα για τις μέρες Ό,τι θέλετε θα πρέπει να απευθύνετε στη γραμματεία. Επίσης, σήμερα συνδέσουμε εδώ, αλλά προσέξτε, αύριο, αύριο θα συνδυάσουμε σε αυτό το κτίριο, στον 5ο όροφο, στην αίθουσα 5β001. Οπότε μην ξεχάσετε να πάρετε τα έγγραφα μαζί σας επίσης ο κανονισμό για τι γενικευμένες προτιμήσει όπου εγκρίθηκε από την Ολομέλεια των Ιόνιων ε, έχει αναθεωρηθεί από τη νομική υπηρεσία σύμφωνα με τη διάταξη 216 αποτελεί το διορθωτικό κείμενο και έχουμε κάποιε αλλαγέ στο κείμενο οι οποίες ε, είναι γλωσσικού χαρακτήρα δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα και θα επικυρωθεί αυτή, αυτό το διορθωτικό έγγραφο το Σεπτέμβριο στην Ολομέλεια. Επίσης, Έχουμε δύο νέα μέλη, τα καλωσορίζουμε. Α, όχι, δεν ήρθαν ακόμα. Κυρία Νόρα Μπέρα, που αντικαθιστά τον κύριο Αμπά και τον κύριο Χένρι Βέμπερ, που αντικαθιστά τον κύριο Αρίφ. Α, δεν το ξέρατε. Item 4. Πάμε στο σημείο υπεριθμών 4. Πρόοδος των τριμερών διαπραγματεύσεων σε σχέση με το πολιετές, δημοσιονομικό πλαίσιο και το σχετικό κανονισμό. Μάρτιν, δικό σου θέμα είναι. το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αξιότιμοι συνάδελφοι, Πολύ σύντομα μόνο θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάτι. Πρόκειται για τον τριμερή διάλογο. για το σχέδιο κανονισμού που αφορά το χρηματοοικονομικό πλαίσιο για τρίτες χώρες. Είχαμε δύο είδη συναντήσεις των τριμερών αυτών διαλόγων στις διαπραγματεύσεις υπό την Δανέζικη Δανική Προεδρία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Προεδρία αυτή της Δανίας για το επικοδομητικό πνεύμα και την αρρωγή που μας παρέσχουν σε αυτές τις συνεδριάσεις. Είχαμε τη συνεδρίαση στις 4 Ιουνίου, είχαμε ανταλλαγή, ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων στις βασικές θεμελιώδεις αρχές και τοποθετήσεις των θεσμικών οργάνων Επίσης παρουσιάσαμε σε σχέση με το Ευρωκοινοβούλιο αρχές σύμφωνα με το ψήφισμά μας στοιχεία σε σχέση με το ψήφισμα που εγκρίναμε πρόσφατα και στις 28 μετά την 4η Ιουνίου στις 28 Ιουνίου συναντηθήκαμε για δεύτερη φορά εκεί εξετάσαμε λεπτομέρειες σε μεγαλύτερο βάθος εξετάστηκαν ε, οι θέσεις αναάρθρο σε σχέση με το σχέδιο κανονισμού και είχαμε μια πραγματικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Πολλά απομένουν σίγουρα ακόμα και πρέπει να γίνουν γιατί δεν πετύχαμε να διευθετήσουμε πολλά από τα επίμαχα θέματα σε σχέση με αυτό το θέμα. Θα το προσπαθήσουμε να το πετύχουμε στην επόμενη συνεδρίασή μας. Η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου. Ήδη φυσικά έχει αποφασιστεί ότι θα προεδρεύει η Κυπριακή Προεδρία όπως είναι φυσικό. Και στην επόμενη συνάντησή μας προσβλέπουμε στο να μπορέσουμε να πετύχουμε ένα αμοιβαία αποδεκτό συμβιβασμό και να καταφέρουμε να επιλύσουμε τα περισσότερα επίμαχα θέματα σε σχέση με το σχέδιο κανονισμού. Φυσικά ως Ευρωκοινοβούλιο έχουμε στεναρές θέσεις στις τοποθετήσεις μας επί πολλών θεμάτων και αναμένουμε ότι θα μπορέσουμε να επιτύχουμε συμφωνία με τους συναδέλφους μας των άλλων θεσμικών οργάνων επ' αυτών των θέσεων. Σε <clears throat> ευχαριστούμε. Θέλει κάποιος το λόγο από τους συναδέλφους. Όχι. Καλώς. Τώρα προχωρούμε. Όσον αφορά τις, ε, αυτές τις ε, αυτόνομες προτιμησιακές ρυθμίσεις που είπαμε στην εισαγωγή, έχουμε τριμερή διάλογο, ο οποίος έγινε στις 14 ε, έκτου. Είστε Ελλάδα τις αναφερμένες προτάσεις από την Προεδρία. Ο πρόεδρος σας ε, θα ε, παρασκευή και θα μιλήσει σήμερα κάποια στιγμή ε, εδώ θα μας πει τι έγινε στον τριμμένο διάλογο και όπως είπαμε στην εισαγωγή εάν προκύψει κάποια λύση τότε θα γίνει αύριο η σχετική ψηφορία. Καταρχήν έχει πει ναι το Συμβουλίο αλλά θα πρέπει να χτενίσουμε ε, τις λεπτομέρειες για να δούμε αν όλα γίνανε όπως πρέπει. Το 5 αναβάλλεται. Και πάμε στο 6. Ενδιάμεση έκθεση εν ώψη της θετικής έκβασης της διαδικασίας έγκρισης του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Σάιτ Καμάλ είναι ο εισηγητής. Ε, θα έπρεπε να σας μιλήσω εγώ, αλλά δεν μου έχουν δώσει ακόμη τις σημειώσεις. Μήπως κάποιος θέλει κάτι να πει σε αυτό το θέμα. Ο κύριος Καμάλ δεν είναι εδώ, ούτε θα είναι εδώ. Ποιοι είναι οι σκιώδεις. Η Επιτροπή θα λάβει το λόγο. Ο το λόγο μπορεί να σχολιάσει και θα θεωρηθεί ότι αυτό είναι μια πρώτη συζήτηση και ο κύριος Καμάλα οφείλει να το δεχθεί. Και τώρα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριος Λιπόντε. Έρχονται συναδέλφοι, δεν, δεν είναι ακόμη εδώ. Πάντως είναι καθοδόν. on that note, then, if the, if you let... Πέστε μου, όταν έχουν έρθει και θα του δώσουμε το λόγο. Οπότε, αν δεν έχει αντίρρηση, προχωρούμε πάνω στο υπαριθμό 7. Να, αυτό γίνεται όταν κανένα αρχίζει την ώρα του. Δεν έχουν έρθει αυτοί που πρέπει διαδικασίε εφαρμογή τη Συμφωνία Σταθεροποίηση και Σύνδεση Ευρωπαϊκή Ένωση Σερβία και Προσωρινή Συμφωνία Σερβία και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μόλι έφτασα, έχω την ευκαιρία να παρουσιάσω κάποια θέματα. Πρόκειται για μια έκθεση για τον κανονισμό εφαρμογής όσον αφορά τη Συμφωνία σταθεροποίηση ΕΕ και Σερβίας Σταθεροποίηση και εταιρική Σχέση. Η προσωρινή αυτή συμφωνία στις 29 Απριλίου υπεγράφει και δεν άρχισε ακόμα να ισχύει επειδή πρέπει φυσικά να επικυρωθεί από τα κράτη-μέλη πρώτα. Υφίσταται μια προσωρινή συμφωνία σε σχέση με το συνολικό τμήμα της ε, συμφωνίας αυτής και προτείνει αυτό τον εφαρμοστικό κανονισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προσωρινή αυτή μεταβατική συμφωνία. Βρισκόμαστε σε παρόμοια κατάσταση όπως με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, την Κροατία, Βοσνία, Ζεγοβίνη, Μαυροβούνια κτλ. εφαρμόζοντας αυτές τις διατάξεις και με τις διαδικασίες ε, επιτροπολογίας ε, και σε σχέση με τις προτάσεις Omnibus 1 Ήδη από πλευρά Κοινοβουλίου έχετε ασχοληθεί με αυτά τα θέματα. Ήδη τον Μάρτιο εφέτος σε σχέση με το Omnibus 1 για να διατηρήσουμε την ίδια γραμμή πορείας και να διασφαλιστεί η συνεκτικότητα και συνέχεια στην, στις τοποθετήσεις προτείνω τις αλλαγές αυτές που έχουν ήδη εγκριθεί στο Omnibus 1. Αφορούν αυτές οι μεταβολές διαδικασίες συμβουλευτικές σε περίπτωση κατεπηγόντων και τη διευκόλυνση της ε, εκμετάλλευσης της χρήσης ε, της, ε, των γραπτών εγγράφων διαδικασιών. Κάποια σχόλια λοιπόν σχετικά, Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η Συμφωνία Εταιρική Σχέσης και Σταθερότητα στοχεύει να δημιουργήσει ένα χώρο ελευθέρου εμπορίου μεταξύ της ΕΕ και της συνολικής περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων. Τον Φεβρουάριο 2010 είχαμε μια προσωρινή συμφωνία που άρχισε να ισχύει μεταξύ ΕΕ και Σερβίας. Χωρίς όμως εφαρμοστικό κανονισμό δεν μπορεί να υλοποιηθεί να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία. Εξακολουθεί να επωφελείται από αυτόνομη αυτόνομο καθεστώς που της έχει αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι προς το συμφέρον μας λοιπόν να αρχίσει γοργά να ισχύει. Είναι δηλαδή προς όφελος όλων να έχουμε μια ταχεία υλοποίηση και εφαρμογή αυτού του κανονισμού. Φυσικά εξαρτάται αυτή η έκβαση του κανονισμού αυτού από την έκβαση των προτάσεων Omnibus 1. Γνωρίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές δεν έχουν αρχίσει ακόμα. Λόγω της περιπλοκότητας του ζητήματος το Συμβούλιο δεν κατάφερε να συμφωνήσει ακόμα σε σχέση με την εντολή, διαπραγματευτική εντολή. Γι' αυτό ζητώ από τη νέα Προεδρία του Συμβουλίου, την Κυπριακή Προεδρία, να αυξήσει τις προσπάθειες για αυτό το στόχο, να απελευθερωθούν, να ξεπαγώσουν όλα τα χαρτοφυλάκια σε σχέση και με τις διεργασίες επιτροπολογίας. Έχουν ήδη περάσει δυόμιση χρόνια από τότε που άρχισε να ισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας. Πιστεύω ότι ήρθε ήδη η χρονική στιγμή πια να γίνουν αυτές οι προσαρμογές ώστε να προσαρμοστούν οι διατάξεις όσον αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνας ακολουθώντας την θέση της Κοινοβουλευτικής μας Επιτροπής που προηγούμενα είχε εκφραστεί μετά από διάφορες συζητήσεις και διαβουλεύσεις για προσαρμογές σε σχέση με τα θέματα επιτροπολογίας. Ελπίζω θα με υποστηρίξουν σε αυτό το αίτημα οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ. Κύριε Σούστα παρακαλώ. Ο κύριος Σούστα. Ε, Ευχαριστώ. Εγώ αντικαθιστώ τη συνάδελφο Κοπά, η οποία είναι η σκιώδη συγγήτρια. Εγώ δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω στο κατά πόσο είναι σημαντική αυτή η συμφωνία σταθεροποίησης με τη Σερβία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ολοκληρώσουμε την διαδικασία προσχώρησης των Βαλκανίων φυσικά με τα κατάλληλα χρονοδιογράμματα και τρόπους. Ενισχύουμε τις εμπορικές σχέσεις με τη Σερβία, και τις ε, διμερείς ε, σχέσεις μεταξύ Ένωσης και Σερβίας. Όπως υπογραμμίζει και η συνάδελφος Κοπά, θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία όπως υπογραμμίστηκε και στο συμπερασματικό τμήμα της ε, τοποθέτησης του εισηγητή. Υπάρχουν ε, τα προβλήματα που συνδέονται με την καθυστέρηση έγκρισης αυτού του νέου κανονισμού. Υποστηρίζοντας εμείς τις τροπολογίες που πάνε προς την σωστή κατεύθυνση έτσι όπως προτείνονται από τον εισηγητή, θεωρούμε ότι και η Προεδρία πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της ούτως ώστε να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο το οποίο και σκόπιμο να είναι αλλά και υποστηρίξιμο από την πλειοψηφία του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ματσίν, θες κάτι από τους φιλελεύθερους? Ο Φράνσις Κέλλο. Ή Φράνσις Ευχαριστώ και εγώ σύντομα να πω ότι εμεί οι πράσινοι υποστηρίζουμε πλήρω αυτή την προσέγγιση και είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβουλίο να ασκήσει αυτέ τι ε, αρμοδιότητε του και να μην υπαναχωρήσει. Μπορούμε να υποστηρίξουμε απόλυτα την έκθεσή σα. Ε, Ευχαριστούμε. Κάποιο από την Επιτροπή παρίσταται. Ο κύριο Κάνερ, ίσω, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει παρατηρήσει σε αυτή τη φάση, δεν έχει σχόλια. Ευχαριστώ. Okay. Jules, you want to come back? <laughs> Εντάξει, εσείς, ε, Jules, θέλετε να επανέλθετε. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω για τις παρατηρήσεις. Έτσι θα συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Right. Uh, deadline for amendment. Εντάξει, προθεσμία για τις τροπολογίες 20 Ιουλίου, 12 το μεσημέρι. Ευχαριστώ. Και έτσι θα επανέλθουμε τώρα στην ε, άλλη έκθεση. Έχουμε τώρα κάποιον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό, για την έκθεση Καμάλ. Το όνομά σας εσάς. Λουμποντέ, ε? μάλιστα. <laughs> Θα ήθελα να κάνω ένα γενικότερο σχόλιο για τη διασύνδεση μεταξύ της πολιτικής εμπορίου και την ανάγκη για πρόσθετα κονδύλια για τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Όπως γνωρίζετε έχουμε ένα φιλόδοξο πλαίσιο για την ημερήσια διάταξη, για το θεματολόγιο, για τις διαπραγματεύσεις που θα πρέπει να αρχίσουν και να συνεχιστούν. Δεδομένης της χρηματοοικονομικής ε, συγκυρίας, το εμπόριο έχει θεμελιώδη σημασία για την ανάκαμψη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα όσον αφορά τη, τη σημερινή οικονομική επιβράδυνση, την κρίση του ευρώ και μια μειωμένη ζήτηση από οικονομικής πλευράς. Προφανώς δεν θα εξαφανιστεί, δεν θα απαλληφθεί αυτή η κρίση και αυτό καθιστά ακόμα πιο σημαντικό για μας την πολιτική εμπορίου και επενδύσεων να την χρησιμοποιήσουμε για να προαχθούν οι στόχοι για την οικονομική σταθερότητα, ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης. Για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρξουν τα αναγκαία κονδύλια. Αυτό που θέλουμε να στείλουμε ως μήνυμα σε εσά σήμερα το πρωί είναι ότι έχει υποβληθεί μια πρόταση για πρόσθετα κονδυλία όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχει δύο πτυχές αυτή η πρόταση. Πρώτον, όσον αφορά την ανάπτυξη και μετάθεση και χρήση στελεχών και θέσεων σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρακολούθηση και την επιβολή αυτών των πολιτικών, μπορούμε να απελευθερώσουμε κονδύλια και να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια όταν απελευθερωθούν για να χρησιμοποιηθούν εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο και δεύτερον για μια φιλόδοξη ημερήσια διάταξη που έχουμε πολλές φορές συζητήσει μαζί σας και χρειάζονται αυτά τα κονδύλια. Αυτές οι διαπραγματεύσεις ε, εκτιλήσονται εκ παραλίλου, διαρκούν πολλές φορές δύο ή τρία χρόνια και υπάρχουν δυσκολίες με τα κονδύλια που έχουμε και πρέπει αυτά να είναι περισσότερα. Το μήνυμα που θέλουμε να σας στείλουμε είναι, θέλουμε σας στείλουμε είναι ότι εκτιμούμε ιδιαίτερα την υποστήριξη του Κοινοβουλίου για να υπάρξουν πρόσθετα κονδύλια για τη γενική μας διεύθυνση. Ευχαριστώ. Um, uh, Δύο μιλητές έχουν ζητήσει τον λόγο. Μπέρντε εσείς Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι είναι και σκόπιμο και λογικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πάρει περισσότερα κονδύλια, μια και τα χρειάζεται. Μια και επειδή έχουμε τις τροποποιήσεις, τις μεταβολές της συνθήκης Λισαβόνας και τα δίκανης αυτά, τα στελέχη και τα άτομα στην ε, Γενική Διεύθυνση έχουν παραμείνει τα ίδια και υπάρχει μεγάλη διαφορά που πρέπει να καλυφθεί σε σχέση με τις ανάγκες. Ερώτηση, τι γίνεται με τις δραστηριότητες της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίου στον εξωτερικό τομέα για το εξωτερικό εμπόριο. Δεν επαρκεί μόνο να έχουμε συμφωνίες εμπορικές με κάποιες χώρες Πρέπει επίσης στη συνέχεια και στις πρεσβείες μας στο εξωτερικό να έχουμε εμπορικούς ακολούθους που θα βρίσκονται εκεί για να παρακολουθούν αυτά τα θέματα, που θα διευκολύνουν και θα υποστηρίζουν τις ευρωπαϊκές βιομηχανίες για να βρίσκουν ευκαιρίες διείσδυσης στις αγορές των άλλων αυτών χωρών. Αυτό το έχετε σκεφτεί στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις αρμόδιες αυτές πρεσβείες στο εξωτερικό, με τη διπλωματική υπηρεσία να υπάρχουν και ακόλουθοι εμπορικοί ώστε επιτόπου οι θετικές επιπτώσεις σε σχέση με τις συμφωνίες εμπορίου να μπορούν να υλοποιηθούν. Okay, thanks. Εσείς λοιπόν, κάπως ε, με ξενίζει αυτό. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Αυτή η έκθεση του κυρίου Καμάρ θα αφορά μόνο πρόσθετα στελέχη για τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Όπως φαίνεται τώρα υπάρχουν και άλλες πτυχές σε αυτή την έκθεση που έχουν ενδιαφέρον δεν είμαι κατά του να υπάρχουν πρόσθετα στελέχη για τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και για άλλε γενικέ διευθύνσει που έχουν πρόσθετο έργο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά αυτό δεν μα βοηθάει ουσιαστικά. Αν δείτε την ημερήσια διάταξη τη Επιτροπή ΣΥΝΤΑ, υπάρχουν τόσα πολλά σημεία που υπάρχουν δυσκολίε Δηλαδή να εξοικειωνόμαστε με όλα αυτά και να μπορούμε με αυτούς τους ρυθμούς να τα καλύψουμε. Ποιος θα μπορέσει να τα καλύψει όλα αυτά το Ευρωκοινοβούλιο. Πώς θα κάνουμε σωστή δουλειά όταν θα αυξάνονται οι ρυθμοί και θα γίνονται όλο και πιο γοργοί, ταχύτεροι και ποιος θα τα παρακολουθεί και θα τα καλύπτει αυτά. Ήδη τώρα είναι δύσκολη η δουλειά μας. Το να επιταχύνουμε τα πράγματα δεν νομίζω ότι θα βοηθούσε πολύ. Μπορείτε να εξειδικεύσετε πώς το βλέπετε και τι θεωρείτε ότι είναι κατεπήγοντες τομείς. Τι θα γίνει σε σχέση με αυτά με αυτούς, με τα στελέχη και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι μας βοηθά συνολικά στις ε, κοινοβουλευτικές διεργασίες κάτι. Thank Σας ευχαριστώ κύριος Μέρφυ. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα πώς χρησιμοποιούμε τα κονδύλια μας, για ποιους στόχους. Δεν είναι μόνο να ζητάμε περισσότερα κονδύλια. Πώς χρησιμοποιούνται είναι σημαντικό. Ένα από τα στοιχεία είναι ότι οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και ο τρόπος με τον οποίο ακολουθείται η πολιτική στην Ευρώπη, η πολιτική λιτότητα καταστρέφει τις εσωτερικές αγορές. Και έτσι οι εξαγωγές φαίνεται να, υπάρχουν, να δίνουν μια δικλίδα ασφαλείας. Το διεθνές εμπόριο παίρνει όλο και μεγαλύτερη σημασία δεν είναι όμως λύση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, στην Ευρώπη και για τους εργαζόμενους στην Ευρώπη γενικότερα, γιατί η πολιτική λιτότητας έχει και θα έχει αρνητικές επιπτώσεις γενικά στην παγκόσμια οικονομία και δεν υπάρχει διαφυγή. Το να έχουμε περισσότερα κονδύλια, να ακολουθούμε την ίδια νεοφιλελεύθερη ημερήσια διάταξη με το ίδιο θεματολόγιο και τι ίδιε συμφωνίε εμπορίου, δεν θα συμφωνούσαμε με κάτι τέτοιο. Ένα άλλο θέμα είναι από πού προέρχονται αυτά τα κονδύλια. Δεν έχει νόημα το εμπόριο και ακόμα πώς να το πω, εξειδικευμένες ε, πτυχές του εμπορίου να υποκαθιστούν την αναπτυξιακή βοήθεια και την πολιτική μας γι' αυτό. Thank Σας ευχαριστώ. Για διαδικαστικό θέμα μόνο. Βλέποντας όσα έχουν σημειωθεί σε σχέση με τον κύριο Καμάρ, έχει αλλάξει η προθεσμία από τον Οκτώβριο στο Σεπτέμβριο, έχει επισπευστεί σε σχέση με τη, τα θέματα του προϋπολογισμού. Ξέρει κανείς ε, γιατί έγινε αυτό, γιατί επισπεύστηκε αυτή η ημερομηνία. Επανέρχομαι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Κάνουμε λόγο για το πόσο γρήγορα, πόσο γοργά θα περάσει αυτό το θέμα. Και το έχετε επισπεύσει κιόλα στην ημερομηνία, παρακαλώ. Η Επιτροπή, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, Ας ξεκινήσω ίσως με τη δεύτερη ερώτηση για τις ανάγκες που υπάρχουν, διότι προφανώς πράγματι κάναμε μια πολύ προσεκτική ανάλυση και αξιολόγηση, αναθέση και για κάθε στέλεχος για τις ανάγκες για αυτές τις διαπραγματεύσεις και έχουμε συνειδητοποιήσει πλήρως ε, το κλίμα, τον περίγυρο λιτότητας και την δέσμευση μειώσεων και τα λοιπά που έχει αναλυφθεί. Όπως είπα είναι γνωστό σε σχέση με τις φιλο, τους φιλόδοξους στόχους για την ημερήσια διάταξη για τα θέματα εμπορίου. Με 11 περιφέρειες και οι χώρες έχουμε τέτοιες διαπραγματεύσεις και δυνατότητες να ανοίξουν και περαιτέρω. Και μέχρι το 2013 θα έχουμε 13 επιπρόσθετες άλλες διαπραγματεύσεις που θα διπλασιάσουν τα όσα τεκταίνονται αυτή τη στιγμή. Το δεύτερο στοιχείο φυσικά είναι το να διαπραγματευτεί κανείς μια συμφωνία είναι μια πτυχή αυτών που κάνουμε. Όπως είδαμε όμως, η φύση αυτών των συμφωνιών έχει αλλάξει εντωμεταξύ. Έχουμε μετακινηθεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο όχι μόνο συζητήσεων για θέματα μειώσεων των δασμών και των δασμολογικών θεμάτων, αλλά περνώντας και σε πιο κανονιστικά θέματα από πλευράς ρυθμίσεων και διατάξεων. Χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια για να επικεντρωθούμε στην υλοποίηση και συμμόρφωση με αυτές τις συμφωνίες και διατάξεις που έχουμε διαπραγματευτεί και υπογράψει με αυτές τις χώρες. Είναι όλο και πιο δύσκολο σε χώρες όπου υπάρχει αύξηση του προστατευτισμού και των μέτρων προστατευτισμού Βραζιλία, Αργεντινή, Ρωσία να κάνουμε παρακολούθηση και εποπτεία σε σχέση με όλα αυτά και την εφαρμογή τους. Χρειάζονται περισσότερα κονδύλια, χρειάζονται γλωσσικές δεξιότητες και ικανότητες, συγκεκριμένα προφίλ, δηλαδή συγκεκριμένες δεξιότητες και ικανότητες τελεχών. Έχουμε και νέες ε, αρμοδιότητες όσον αφορά τις επενδύσεις που απορρέουν από τις συνθήκες Λισαβόνας. Και αυτό είναι ένα τομέα που θα θέλαμε να αναπτύξουμε σε αυτόν τις δραστηριότητε μας. Υπάρχει τεράστιο δυναμικό δυναμικό και για μικρές και για μεγαλύτερες και μεγάλες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Εκεί θα χρειαζόμαστε πάλι πρόσθετα κονδύλια σε σύγκριση με αυτά που έχουμε σήμερα. Όπως είπα κάναμε μια εξειδικευμένη προσεκτική ανάλυση αυτών που υπάρχουν και έχουμε ως ανάγκες επιπλέον βασιζόμενοι σε διάφορα σενάρια πάντα με βάση την ταχύτητα και τον ρυθμό που θα ακολουθείτε με βάση τις διαπραγματεύσεις. Είμαστε ε, στη διάθεσή σας για περισσότερες λεπτομέρειες. Σε σχέση με το τι γίνεται στο γενικό στρατηγείο, στο κέντρο και στις περιφέρειες, στις χώρες, στις αντιπροσωπείες και στα κράτη-μέλη και φυσικά στις πρεσβείες επιτόπου, για εκπροσώπηση έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για να υπάρξει καλύτερη διάρθρωση αυτών των, ε, αυτής της εκπροσώπησης και σε, καλές, ε, σε καλή σχέση με τις χώρες και τα, τις πρεσβείες. Ιδιαίτερα για αυτές τις μεγάλες αναδυόμενες αγορές για παράδειγμα. Δημιουργήσαμε ομάδες πρόσβασης στην αγορά, πελασιμότητας για να εξεταστούν τα προσκόμματα και τα εμπόδια επιτόπου να δούμε τι γίνεται σε σχέση με τις επιχειρήσεις, ποια εμπόδια αντιμετωπίζουν, ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν για να αρθούν, να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια. Και όλα αυτά σε ένα συσχετισμό και συνεργασία επικοδομητικό και γόνιμο. Επίσης εσωτερικά προβληματιζόμαστε για το πώς θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτά τα κονδύλια από πλευρά πλευράς αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια έκθεση θα υποβληθεί όσον αφορά το workload assessment, δηλαδή την αξιολόγηση του φόρτου εργασίας και το τι πρέπει να γίνει σε σχέση με τις αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παγκόσμια. Στόχος είναι να μετατεθεί και να να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες το προσωπικό, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ανάγκες των αναδυόμενων χωρών και αναδυόμενων οικονομιών. Δεύτερο, και εκεί πάλι σε σχέση με το τμήμα της Γενικής διεύθυνση Εμπορίου, ζητήσαμε μια μετριοπαθή αύξηση στελεχών σε κάποιες αντιπροσωπείες διότι σε σχέση με ένα δίκτυο 153 τέτοιων αντιπροσωπιών παγκόσμια δυστυχώς υπάρχουν στελέχη επαρκή μόνο σε ένα τρίτο ουσιαστικά ε, σε αθρές γραμμές για τις αντιπροσωπείες. Υπάρχουν λοιπόν πολύ μεγάλες ανάγκες. Δεν υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι για το εμπόριο που να μπορούν να καλύψουν ε, αυτές τις πρόσθετες ανάγκες είτε για την πρόσβαση στις αγορές είτε για κανονιστικά θέματα και ε, διατάξεις και κανονισμούς. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτά τα πράγματα όχι μόνο στο κεντρικό μας, στο κέντρο μας στις Βρυξέλλες αλλά και στις αντιπροσωπείες. Εργαζόμαστε πάρα πολύ στενά λοιπόν και με τα κράτη-μέλη και τις πρεσβείες για να καλυφθούν αυτά τα κενά. Ευχαριστώ. Μόλις τώρα μου είπαν Θα σαν τη λίστα τώρα με αυτού οι οποίοι ενδιαφέρονται για το θέμα του κ. Καμάλ. Για, έχουμε τι τέσσερι ερωτήσει που λέτε πέρα. Πρώτα-πρώτα η σημερινή αρχιτεκτονική. Ε, αυτή, ε, ε, αν καλύπτει τους ε, στόχους της εμπορικής πολιτικής για την οικονομική συνεργασία. Θεωρείτε ότι αυτοί οι στόχοι εξυπηρετούνται από αυτές τις δράσεις όσον αφορά τα ε, μέσα πολιτική γενική δράση. Επίση, ε, αυτά τα οποία έχει πει για τον τέταρτο τίτλο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά ε, αυτό σαν πρικοδότηση είναι εντάξει. Τρίτον, τι γίνεται με τα εξωτερικά εργαλεία, θεωρείτε ότι υπάρχει η σωστή ισορροπία, για αν όχι γιατί. Και τέταρτο και σημαντικό, έχουμε αρκετή συνέπεια μεταξύ των μέσων πολιτικής των εργαλείων και της εφαρμογής. Πιστεύετε ότι ε, οι διοικητικές δαπάνες οι οποίες έχουν διατεθεί είναι ε, αρκετές επαρκείς, επίσης από πλευράς διαδικαστικής η ψήφιση θα γίνει 10 και 11 δεκάτου αυτό σημαίνει ότι πιεζόμαστε πάρα πολύ ούτως ώστε να έχουμε έτοιμη την γνωμοδότηση εγκαίρως και Έχουμε αυτή την ψήφιση. Από εμά θα γίνει μεταξύ 17 ή 18, ή 18 Σεπτεμβρίου και όχι 10-11 Οκτωβρίου. Άρα ένα μήνα πριν. Επομένω θα πρέπει να έχουμε τα κείμενα, τις μεταφράσεις. Αυτό βέβαια ε, έχει ξεφύγει, ε, δεν είναι θέμα δικό μας, τώρα γιατί έχει γίνει αυτή η αλλαγή, δεν ξέρω, Πώ το είπατε. Τι μέρα. 5 ενάτου είναι η για τις τροπολογίες. Ναι, όλοι θα ειδοποιηθείτε και έτσι ε, θα είναι όλα έτοιμα εγκαίρως. Πότε θα λάβουμε τα έγγραφα, λέει ο κ. Λάγκη, από τον κύριο Καμάλ. Πώς να κάνουμε τροπολογίες χωρίς τα έγγραφα. Τέλος του μήνα αυτού. Okay. Yeah. This who's uh, the... Establishing a θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για συνεργασία. Να δούμε τώρα τι έχουμε τα χρηματοδοτικά μέσα για ανάπτυξη και συνεργασία. Φορά ένα νέο κανονισμό 2014-2020. Η Επιτροπή Ανάπτυξη είναι κυρίω ε, αρμοδία επιτροπή και τώρα ο Χέλμουντ έχει το λόγο. Θέλει το λόγο. Χέλμουντ Σόλτ. Ήδη τα έχουμε συζητήσει όσον αφορά ε, αυτό το θέμα την τελευταία μας συνεδρίαση. Και εγώ είχα υποβάλει κάποιες προτάσεις, σας είχα πει τι θέλω να κάνουμε για αυτή την γνωμοδότηση, οπότε απλώς σας τονίζω στην αρχή ότι υπήρξε η ευκαιρία να επεξεργαστούμε μαζί με άλλες επιτροπές μια γενική γραμμή για το περιεχόμενο, τη δομή και το βεληνικές αυτό σε σχέση και με την ε, ΑΦΕΤ και σε σχέση με τις τροπολογίες προσπάθησα να συνεργαστώ με την Επιτροπή για να ευθυγραμμιστούμε. Η Επιτροπή Ανάπτυξης την ε, περασμένη εβδομάδα μας συνάντησε, κάναμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και είπαμε ποιες είναι οι νέες προτάσεις για το χρηματοδοτικό μέσο, DCI. Θέλουμε να υπάρχει απλούστευση να φρεμιστούμε με τους εταίρους μας άλλες χώρες, να υπάρχει διαφοροποίηση ανά χώρα και ανά τομέα. Μέσα τόσο έχουμε πάντως 200 τροπολογίες. να τι κάναμε εμείς εδώ. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω τους και οδησηγητές. Με τα τελευταία μας συζήτηση ξεκινήσαμε λοιπόν την τελική ευθεία για την επεξεργασία αυτής της γνωμοδότησης και ελπίζω ότι όπως πήγαμε μέχρι τώρα θα, προχωρήσουμε σωστά μετά τη σημερινή συνάντηση. Επίσης, σας τονίζω τα εξής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο γενικώ ε, ισχύει. Θα πρέπει να δούμε πώς θα καθορίσουμε τους βασικούς στόχους της αντισιακής συνεργασίας. για τον μηχανισμό χρηματοδότηση 2014-2020 και για άλλη μια φορά. Σα τονίζω αυτό το οποίο έκανε και την τελευταία φορά ότι ο στόχος αυτός της εμπλησιακής πολιτικής παραμένει ούτως ώστε να μπορέσουμε να συμβάλλουμε στην εκρίζωση της φτώχειας ακριβώς όπως ορίζει και συνθήκη την Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να συζητούν και στην Επιτροπή ε, Διεθνούς Εμπορίου είναι μια πρόκληση, θα πρέπει να εστιάσουμε προσοχή μας και να μην το ξεχνούμε κάθε φορά που ασχολούμεθα με το σχέδιο γνωμοδότησης το δικό μου. Να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις ε, ελαφρές τροποποίησεις που έχει προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το μηχανισμό χρηματοδότησης, το DCI, ούτως ώστε να ευθυγραμμιστούμε με τις ε, σημερινές αντισιακές πολιτικές. Αλλά για να βελτιώσουμε και αυτή την προσέγγιση, την πρότασή μου πρότεινα να δούμε τι θα γίνει με το παράδειγμα 5, ούτως ώστε να, να αλλάξει το, το κείμενο το νομοθετικό. Επίσης έτσι θέλουμε μια διαφοροποιημένη προσέγγιση, συμφωνεί και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να εστιάσουμε προσοχή μας σε χώρες και σε περιφέρειες. Πάντως, θα πρέπει να δούμε τι ανάγκες υπάρχουν ακριβώς σε στενή συνεργασία με τις χώρες με τις οποίες θα έρθουμε σε επαφή Οπότε, αυτά να σου δούμε στο συμπέρασμα ότι κάπως υπερέβαλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάποιες χώρες άφησε απ' έξω από την ε, συνεργασία, την αναπτυξιακή. Άρα θα πρέπει τώρα να επανεντάξουμε στο, στην πολιτική μας αυτή κάποιες χώρες, ε, στο παράδειγμα υπαριθμών 3, κυρίως χώρες της Λατινικής Αμερικής, να τις ξαναβάλουμε στον κατάλογο των επιλέξιμων χωρών. Επίσης, να δούμε πώ θα έχουμε το, ένα αποτελεσματικό μηχανισμό χρηματοδότησης. Πάντως ε, δεν θα πρέπει με την ευελιξία να απεμπολίσουμε τις ε, κοινοβουλευτικές μας υποχρεώσεις γιατί ακόμα και μια μικρή χώρα ε, χρειάζεται τα έστω λίγα χρήματα. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα ποσό που να θεωρηθεί ότι είναι πάρα πολύ μικρό. Όλα τα χρειάζονται, όλα τα ποσά χρειάζονται σε κάποιες, σε... οι χώρες αυτές. Και είπαμε για αυτή τη λευκή πενταγή ε, που να πρέπει να φτάσει στο 60% και θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο αποδέχεται αυτή την πρόταση. Επίσης, τονίζουμε ότι θα πρέπει να ξαναεξετάσουμε το τι γίνεται με τους εμπορικούς μας ε, στόχους που θα πρέπει πάντοτε να έχουμε στόχους εμπορικούς που να ευθυγραμμίζονται με τους αναπτυξιακούς στόχους λόγω της αναπτυξιακής συνεργασίας που θέλουμε να έχουμε. Τέλος, χαιρετίζουμε την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περιλάβει εδώ κάποιες νέες γραμμές όπως ας πούμε τη στρατηγική για την Αφρική και αυτό σημαίνει ότι η Αφρική έχει προτεραιότητα σε σχέση με την πολιτική μας για την εκρίζωση της φτώχειας. Αυξήθηκε η σωνική πρικοδότηση και αυτό επίσης μας βρίσκει σύμφωνος σαν κοινοβούλιο. Οπότε με, με όλα αυτά το φθινόπωρο φαντάζομαι το κοινοβούλιο πρόκειται να επιψηφίσει το, το σύνολο των προτάσεων. Όπως σας είπα θα κάνουμε μια συνάντηση επίσης με τους συνεργάτες μας, ε, το διοικητικό προσωπικό του Κοινοβουλίου, τους σκιώδης ηγητές. Κάπως άβολο πάντως ε, είναι το ότι θα πρέπει ε, να συναντηθούμε στις 3 Σεπτεμβρίου με τις διακοπές αμέσως μετά να ψηφίσουμε. Λοιπόν, μήπως γίνεται η γραμματεία να μας βρει ένα άλλο χρονοδιάγραμμα και έτσι να μας δώσει καλύτερα τη δυνατότητα να εξετάσουμε τις τροπολογίες. Ίσως ε, εγγράφως να συνοηθούμε, να βρούμε ε, κάποιες λύσεις, κάποιες συμβαστικές τροπολογίες και έτσι το φθηνό την να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Χέλμοντ, λέει ο πρόεδρο, νομίζω ότι όντω θα, θα έχει κέφια όταν έρθει από τι διακοπέ. Ελπίζω, ελπίζω, λέει ο κύριο Σόλτ. Ναι, αλλά έχουμε κάποιο πρόβλημα. Διότι η αλήθεια είναι ότι ε, η Επιτροπή των Προπολογισμών έφτιαξε αυτό το χρονοδιάγραμμα και νομίζω ότι είναι αδύνατο να αλλάξουν ημερομηνίε. Δεν γίνεται. Θα πρέπει να τηρήσουν αυτό το χρονοδιάγραμμα. Έχουμε βέβαια και μια πράσινη εβδομάδα λίγο πριν αν θέλει κάποιος να έρθει λίγο πιο νωρίς από τις διακοπέ. τότε ναι. Θα, εγώ θα είμαι εδώ στις 31 Οκτωβρίου, λέει ο Χέλμοντ. Να, ε, να δούμε, εσύ θα είσαι. Καλά, ευχαριστώ. Βίγκλερ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Για την κυρία Σαΐφη. Θέλω να μιλήσω ότι δεν μπόρεσε να παραστεί. Τα είπε και ο συγκεκριτή ο κύριο ε, Σόλτζη. μια που χθε συναντήθηκαν τις πιο Οπότε, να σα πω δύο-τρία πράγματα για την συνάδελφο. Πρώτα-πρώτα, κάποιε από τι τροπολογίε θεωρεί ότι δεν είναι αρμοδιότητα της ε, δικής μας Επιτροπής. 30, 31, 32 39 με 50. Πρώτοι αυτές τις τροπολογίες. Αυτές θεωρεί η συνάδελφο ότι είναι εκτό αρμοδιότητα τη Επιτροπής μα. Επίση, συμφωνεί εν μέρη με το περιεχόμενο των τροπολογιών και καταλαβαίνει πού το πάει ο εισηγητής. όπω μα τα εξήγησε πριν, όμω δεν είναι καθόλου βέβαιη ότι αυτή η γνωμοδότηση είναι το κατάλληλο μέρος, το κατάλληλο κείμενο για να καλυφθούν αυτές οι τροπολογίες το 31 που αλλάζει τις επιλέξιμες χώρες κατά, το, κατά τη γνώμη της κυρία Σαΐφη αυτό θα πρέπει να το κάνει η κυρίως αρμόδια επιτροπή στα πλαίσια του τριμερούς διαλόγου ο οποίος όπου να είναι ξεκινάει επίσης ζητά το ΕΛ κάποιες χωστές ψηφοφορίες την τροπολογία υπαριθμών 7 να μείνει ένα τμήμα του αρχικού κειμένου όσον αφορά την αιτιολογική παράγραφο 15. Επίσης, και για το άρθρο 27 επί του άρθρου τροπολογία 27 του άρθρου 14 ε, όσον αφορά την αύξηση ή μείωση των αρχικών ενδεικτικών ε, εκταμιεύσεων σε σχέση με την γενική αυτή διαδικασία. Θεωρούμε ότι η αρχική διατύπωση ε, επιτρέπει αυτού του είδους την διάθεση πόρων για λιγότερο από 20% προτείνει 10%. Λέει λιγότερο του 10% εδώ προτείνεται στην τροπολογία. Η κυρία Σαϊφή λέει ότι δεν είναι θέμα ούτε της ΑΦΕΤ ούτε της ΔΕΒΕ. Ε, και άλλωστε εκεί πέρα οι συγκητές δεν θέλουν να αλλάξει αυτό το κατόφλι. Και η κυρία ε, είπε ότι ε, όποτε θέλει ο συγκητής και οι άλλοι σκιώδες συγκητές ε, να, να την βρουν και να τα συζητήσουν και συμφωνεί με οποιαδήποτε αλλαγή χρονοδιαγράμματος. Ευχαριστώ. Καλημέρα, γιατί μόλις έφτασα, ήμουνα στην Ήτρε. Εγώ είμαι σκιώδης εισηγήτρια για αυτήν την έκθεση στην Ίντα. Και θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά τον εισηγητή για τις τροπολογίες. Το θέμα του διεθνούς εμπορίου δεν είναι και πολύ συγκεκριμένο εδώ. Για να το τοποθετήσουμε σωστά το θέμα πρέπει να δούμε πώς να, περιχαρακώσουμε τις αρμοδιότητες της κάθε επιτροπής. Δεν χρειάζεται λοιπόν να προσπαθεί να μονοπολίσει μία επιτροπή τις αρμοδιότητες για τις, από τις οποίες προκύπτει αυτή η έκθεση. Έχουμε το θέμα του εργασιακού δικαίου, έχουμε το θέμα της παινίας, της βελτίωσης της ποιότητας ζωής και θα ήθελα να βελτιώσουμε και θα παρουσιάσουμε ορισμένες τροπολογίες για το ποια είναι τα κριτήρια που ορίζουν ποιες χώρες μπαίνουν και ποιες χώρες βγαίνουν από αυτή τη λίστα, διότι το ΑΕΠ θεωρούμε ότι θα μπορούσε να αποτελέσει στοιχείο διακρίσεων. Στις χώρες εκείνες που έχουν, υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν συγκεντρωμένο τον πλούτο σε έναν τομέα και πολύ φτώχεια από την άλλη. Ε, επίσης, ε, πρέπει να δούμε τις ε, χώρες που θα βγουν από τη λίστα και θα δούμε ποια θα είναι περίοδος προσαρμογής για να μην έχουν μία διπλή ζημιά και το θέμα του χρονοδιογράμματος θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα σφιγμένο. Δεν χρειάζεται να τρέχουμε πριν ε, από την ώρα μας πάνω από, ε, πριν από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Ξέρετε, το εμπόριο σημαίνει επίσης και ανάπτυξη. Θα έπρεπε λοιπόν να ορίσουμε ένα νέο χρονοδιάγραμμα στην Ολομέλεια του Στρασβούργου και να κοιτάξουμε να καταστήσουμε πιο ευέλικτο το χρονοδιάγραμμα για να έχουμε συμβιβαστικές τροπολογίες και να ψηφίσουμε χωρίς να έχουμε αστεπιασμένοι από το λαιμό και με μια σχετική ξεκούραση. Ευχαριστώ. Τα είπαμε εδώ και ένα χρόνο ότι έτσι θα πρέπει να γίνει για αυτό το χρόνο. Και όπως είπε και ο κύριος Σόλτς για να τα καταφέρει θα γυρίσει μια ροχήτρα από τις διακοπές. Δεν ξέρω αν θα τηρήσει την υποσχεσή του, τέλος πάντων. Φραντσέσκα. Uh, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ για αυτή την έκθεση. Πιστεύω ότι μπορούμε γενικά να την υποστηρίξουμε. Πραγματικά οι περισσότεροι φτωχοί βρίσκονται σε χώρες ε, μεσαίου εισοδήματος ε, και πρέπει αυτό να λαμβάνεται υπόψη. Και ένα μείζον θέμα για την DCI θα είναι να διασφαλιστούν οι εξουσίες του Ευρωκοινοβουλίου όπως ε, έχουν εγγυηθεί και πρέπει να διασφαλίζονται με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Αν δούμε ή βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει ουσιαστικά να έχει κάρτα εν λευκό στο να αποφασίζει τι θα γίνεται με τα τμήματα τα δημοσιονομικά και τα κονδύλια σε σχέση με μια χώρα που δεν θα παίρνει 50, πάνω, από 100, ε, πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ 50 εκατομμύρια ευρώ πιστεύω ότι είναι αρκετά χρήματα και θα πρέπει το Κοινοβούλιο να εμπλέκεται και όχι μόνο η Επιτροπή να αποφασίζει. Και για τη διευρυμένη διαβούλευση με τις χώρε χώρες εταίρους πρέπει να μπορέσουμε να δούμε τις διευρυμένες ε, αρχές ε, ιδιοκτησίας και σε σχέση και με τις πτυχές ε, κλιματικών αλλαγών και όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη και θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να τονίζουμε και εμείς αυτές τις πτυχές και να τονίζουμε και τα εργασιακά δικαιώματα που <clears throat> θα πρέπει να διασφαλίζουμε για κάποιες χώρες που είναι εποφελούμενες από αυτά τα κονδύλια να διασφαλίζονται αυτές οι πτυχές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός όσον αφορά η υποστήριξη που δίνεται σε σχέση με τα θέματα που έχουν κάποια σχέση με το εμπόριο. Αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη και να δούμε ποια άλλα κέντρα βάρους θα προταθούν από την Επιτροπή Ανάπτυξης ε, Συνεργασίας για την Ανάπτυξη. Δεν θα εξεταστούν μόνο οι πτυχές εμπορίου από εκείνους, πράγμα που είναι δική μας δουλειά, πρέπει να αφήσουμε και περιθώριο για εκείνη την Επιτροπή να επικεντρωθεί όπως πρέπει με τον πιο σωστό τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Φραντσέσκα. Άλλος που θέλει να παρέμβει προτού τοποθετηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εντάξει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κύριος Ρένερ, παρακαλώ, ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ και όλα τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής για αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης, ιδιαίτερα και τον κύριο Χέλμουτ Σόλτς Πιστεύουμε ότι είναι μια, ένα σχέδιο έκθεσης που εισάγει και τονίζει, υπογραμμίζει κάποια στοιχεία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε σχέση με όσα αφορούν το εμπόριο και τα συμμεριζόμαστε ως Επιτροπή. Αληθεύει ότι το τελικό προϊόν, ο τελικός κανονισμός που θα εγκριθεί θα πρέπει να είναι καλά ισορροπημένος μεταξύ των διαφορετικών αυτών στοιχείων και για την συνεργασία για την ανάπτυξη και για τα θέματα εμπορίου αλλά και για την ημερήσια διάταξη το θεματολόγιο για αλλαγές και που συζητώνται στο Ευρωκοινοβούλιο. Θα ήθελα να τονίσω κάποια θέματα που μας απασχολούν εμάς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αφορούν ουσιαστικά τρεις άξονες, τρεις τύπους ανησυχίες. Το πρώτο αφορά Αυτές τις διαδικασίες, ε, τις διαδικασίες σε σχέση με τις ε, κατεξοδότηση πράξη και κάποια έγγραφα τα οποία είπαμε ότι θα πρέπει να τροποποιηθούν σύμφωνα με αυτή τη διαδικασία. Βεβαίω αυτό το ζήτημα είναι οριζόντιο. Βέβαια, υπάρχουν και κάποια άλλα ζητήματα που δεν καλύπτονται από αυτό. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε τι θα γίνει για αυτά στι κατευθυντικέ πράξει, οι οποίε ε, ε, θα πρέπει να γίνουν ε, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις διαφοροποίησεις. Γιατί όπως γνωρίζετε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει εδώ να υπάρχει ε, μία διαφοροποίηση σε αυτό το κατάλληλο των 19 χωρών και στη γνωμοδότηση έχουμε πέντε από αυτές τις χώρες οι οποίες είπαμε ότι θα επανενταχθούν ή στον κατάλογο των χωρών που θα καλυφθούν Κολομβία, Κωνσταντίνα, Παναμά, Περού ε, και είπαμε ότι έτσι θα μπορέσουμε να καλύψουμε τους πόρους ούτως ώστε ε, να βοηθήσουμε τις χώρες αυτές και είπαμε επομένως ότι θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Ε, οι χώρες έχουν ακόμα τα προβλήματα, αλλά είπαμε να ε, μην γίνει αυτό με διμερή συνεργασία. Κάτι άλλο το οποίο μας απασχολεί είναι ότι κάποιες από τις προτάσεις αυτές δεν έχουν ευελιξία. Γιατί ένας από τους στόχους της πρότασής μας ήταν να αυξηθεί η δυνατότητα της Ένωσης να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες και στις νέες προκλήσεις. Παράδειγμα, ε, τα παρατήματα 4 και 5 είναι ένας κλειστός κατάλογος από πολιτική επαρρύθμιση και οπότε εγώ έχω ζητήσει ο προγραμματισμός να γίνεται έτσι ούτως ώστε να αντιμετωπίζουν τα πραγματικά προβλήματα. Τώρα έχει κλείσει αυτός ο κατάλογος της δραστηριότητας και για το σχέδιο γνωμοδότησης ε, και φυσικά και για τη δυνατότητα τροποποίησης σε σχέση με το παράτημα όσον αφορά την συνεργασία. Το μη συνεργασία θα παραμένουν ως τμήμα της κανονικής νομοθετικής διαδικασίας. Για αλλαγές πρέπει να ακολουθηθεί κανονική νομική, νομοθετική διαδικασία και για τις μη ουσιώδεις αλλαγές ε, στο, στα προγραμματικά έγγραφα ή για την πρόβλεψη για τα κράτη εκείνα που τα κονδύλια για αυτά είναι 50 εκατομμύρια. Θα θέλω να προσαφηνήσω ότι το γεγονό ότι δεν υπάρχει στρατηγικό έγγραφο δεν σημαίνει ότι δεν θα υποβάλει κάποια στρατηγική η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτέ τι πτυχέ. Θα υπάρχει στο πολιτέ σχέδιο αυτή η παρουσίαση αυτή τη στρατηγική. Δεν χρειάζεται να αντανακλάτε σε δύο ξεχωριστά έγγραφα. Αυτή είναι η πρόταση να πλουστευτεί η διαδικασία για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτέ τι χώρε που έχουν μικρότερα ποσά στη διάθεσή του. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την υπηρεσία εξωτερικής δράσης, την διπλωματική υπηρεσία. Είμαι από την υπηρεσία αυτή και θέλω να σας ευχαριστήσω για το σχέδιο έκθεσης, ειδικά τον κύριο Σόλτς. Πλήρως συμμεριζόμαστε τα σχόλια που έγιναν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον εκπρόσωπό της. Θέλω απλά να υπογραμμίσω ότι πραγματικά σε σχέση με διαφοροποίηση όσον αφορά την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως επεξηγήθηκε από το Χαβιέρ η ιδέα είναι ότι τώρα οι χώρες που έχουν αρκετά κονδύλια για να μπορέσουν να δραστηριοποιηθούν και να αντιμετωπίσουν τα προβλήματά τους δεν χρειάζεται αναγκαία υποχρεωτικά να έχουν διμερή συνεργασία ή να την χάνουν συνδρομή στην διμερή συνεργασία για αυτή την βοήθεια. Αυτό σημαίνει όμως ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλει να οδηγήσει στο να υπάρξει μια νέα μορφή συνεργασίας με αυτές τις χώρες, αλλά να μπορέσουμε να τις βοηθήσουμε περαιτέρω για τα θέματα ανάπτυξης, ιδιαίτερα όσον αφορά το μέσο αναπτυξιακής βοήθειας, που θα μπορούν να υποφελούνται από αυτό αυτές οι χώρες και με την περιφερειακή συνεργασία μεταξύ αυτών των χωρών, ώστε να επιτρέπεται να έχουμε μια γενικότερη στρατηγική σε ένα τέτοιο περιφερειακό πλαίσιο και θα μπορούν τα μέσα και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιούν αυτές οι χώρες να τα αναπτύξουν όπως τα χρειάζονται και το ευρωπαϊκ, τα ευρωπαϊκά μέσα εταιρική σχέσης ή ε, σταθεροποίησης που θα είναι και αυτά σημαντικά μέσα σε αυτό το νέο πλαίσιο εταιρική σχέσης. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Helmut, θέλετε να τοποθετηθείτε εσείς. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα επιστρέφοντας στο χρονοδιάγραμμα. Φυσικά είμαι πρόθυμος και την τελευταία εβδομάδα να είμαι παρόν ώστε με τα άλλα μέλη και τους σκιώδεις εισηγητές είμαστε, είναι ευπρόσδεκτοι να βρούμε ένα συμβιβασμό τότε, να αναζητήσουμε ένα συμβιβασμό. Ίσως αυτό δεν είναι όμως προς το συμφέρον όλων. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε για να αντιμετωπίσουμε αυτό το περίπλοκο θέμα, να βρούμε ένα συμβιβασμό και να έχουμε και ένα πίνακα ψηφοφορίας που θα λαμβάνει υπόψη και τις παρατηρήσεις των σκιωδών εισηγητών. Υπάρχει πρόβλημα και το έχω συνειδητοποιήσει. Θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να βρούμε μια κοινή λύση σε αυτό το πρόβλημα. Δεύτερον, θέλω να ευχαριστήσω για τις παρατηρήσεις που αφορούσαν το ζήτημα του περιεχομένου, της ουσίας, αν είναι αποκλειστικά αρμοδιότητα της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ή και άλλων Κοινοβουλευτικών Επιτροπών. Θα το ξαναδούμε λοιπόν και αυτό και θα το θίξουμε σε σχέση με το άρθρο 27. Και σε σχέση με το άρθρο 27 θα να σας πω ότι βεβαίως ε, για το εξωτερικό εμπόριο και όσον αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Θα πρέπει αυτό να το εξετάσουμε με κάποιο άλλο μηχανισμό, με κάποιο άλλο εργαλείο εξωτερικού εμπορίου και έτσι να καταφέρουμε να έχουμε μια σφαιρική ε, λύση, μια δέσμευση σφαιρική, γενική και νομίζω ότι πάνω σε αυτή τη βάση δούλεψα και οπότε να βρούμε για τις τροπολογίες αυτές μια συμβαστική λύση να μπορέσουμε να προχωρήσουμε αισιόδοξα τις επόμενες εβδομάδες ε, αυτής προσπάθειάς μας για να ολοκληρώσουμε την γνωμοδότησή μας. Και κατά αυτόν τον τρόπο να συμβάλλει η δική μας Επιτροπή σε συνεργασία με την Επιτροπή Ανάπτυξης, τόσο ώστε να ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Επίσης, να δούμε τι θα γίνει με τα παραδείγματα 4 και 5. Και εδώ να ευθυγραμμιστούμε με τις ε, άλλες επιτροπές επί τη βάση των τελικών τοποθετήσεων του Κοινοβουλίου ε, στον τριμερή διάλογο. Το θέμα αυτό με τις κατουσιοδότητες πράξεις δεν είναι καινούριο. Εδώ και Δύο χρόνια ανακύπτει συνέχεια. Γι' αυτό και ελπίζω ότι θα συμφωνήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα συμφωνήσουν οι συνομοθέτες επ' αυτού. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό το μέσο όσον αφορά το ότι θα πρέπει τελικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει τη φωνή του να ακουστεί τώρα. Όσον αφορά τον κατάλογο με τις χώρες Νομίζω ότι και το Συμβούλιο τα ίδια πρεσβεύει. Άρα τελικά νομίζω θα βρεθεί μια λύση. Και ίσως τελικά προσθέτουν ακόμα περισσότερες προσωπικές που εγώ έχω προτείνει αυτά προς το παρόν. Αυτές είναι μου και ελπίζω ότι τελικά θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την γνωμοδότηση μέχρι το Σεπτέμβριο. Θέλουμε λοιπόν, να σε ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Όπως είπαμε, υπάρχει πολύ καιρό για όλους την περίοδο το σχετικό χρονοδιάγραμμα. Άρα έχουμε λοιπόν επόμενη, το επόμενο ορόσημο στις 3 Σεπτεμβρίου, δεν ξέρω μήπως να γενεθλιάσω στη, θα τα πούμε την ΤΕΒΕ στις 18, μήπως το αντί για τις 18 πάμε στις 17 Σεπτεμβρίου, να προσπαθήσουμε. Ίσως αυτό σε βοηθήσει, εσένα και όλους μας. Πάμε στο θέμα υπαριθμών 9, λέει ο Πρόεδρος. Γενικός Προπολισμός Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2013. Έχουμε εδώ συζήτηση από τις γνωμοδότησες και ως συνήθως επ' αυτού ο πάγιος συντάκτης σχεδόν είναι ο Πίτερ, Πίτερ Στάσινη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Για τρίτη φορά συζητούμε αυτό το σχέδιο κειμένο και έχει τώρα την ευκαιρία για τρίτη φορά η Επιτροπή Τεχνικού μπορεί να συζητήσει τα θέματα των προπολογισμών μάλλον του προηγούμενου του 2013, είπαμε ότι εγκρίναμε την εντολή για τον ε, τριμερή διάλογο. Εκεί ορίζονται οι γενικέ προτεραιότητέ μα και κάναμε μετά την ε, πρώτη ανταλλαγή απόψε τον περασμένο μήνα επί του προπολογισμού και τώρα θα δείτε στο σχέδιο του κειμένου μου κάποιε λεπτομερεί προτάσει, ώστε να καλύψουμε τι προτεραιότητε τη Επιτροπή και ταυτόχρονα τι προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το σχέδιο προπολογισμού για το έτο 2013. Και τώρα θα ήθελα με δύο λόγια να σας πω ε, τι, τις συγκεκριμένες μου προτάσεις. Έχω τονίσει το πώς παρά την κρίση δεν θα μειώσουμε τη βασική, τα βασικά κονδύλια του, του βασικού προβλήματο για το εμπόριο. Για όλα μας τα πιλωτικά προγράμματα, για όλες τις προπαρασκευαστικές μας δράσεις. Για όλα αυτά τα οποία θεωρούμε ότι θα αποτελέσουν προστεθεμένη ε, αξία όσον αφορά τις ε, ΜΜΕ και τη διεθνοποίησή τους και τις ε, εμπορικές σχέσεις προς Ανατολάς και προς Νότον. Επίσης, θέλουμε να υπάρχει χρηματοδότηση που να είναι στο ύψος των φιλοδοξιών μας, στο ύψος των στόχων που έχει τάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα αυτά ε, δεν σημαίνουν αύξηση των πληρωμών ή των υποχρεώσεων. Γιατί μιλούμε για ε, το ότι αν είχαμε αυξήσει ε, στον προπολογισμό αυτό, τον εμπορικό, θα ήταν κάτι που θα το καταψήφισε το Συμβούλιο, γιατί ο κόσμο δεν θέλει τέτοια πράγματα, δεν θα, δεν θα μα καταλάβαινε. Ε, δεν θα ήταν ρεαλιστικό. Έτσι κι αλλιώ, τα κονδύλια για το εμπόριο δεν είναι τα πιο αυξημένα στον προπολογισμό. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει όλοι να κάνουμε προσπάθειες για να δούμε ποιες είναι οι προτεραιότητες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να καλύψουμε τους στόχους της Ένωσης και γι' αυτό εγώ θα κατεβάσω ε, κάποιες τροπολογίες επί του δικού μου κειμένου και έτσι θα το επεξεργαστώ, θα το βελτιώσω και κατά αυτόν τον τρόπο επίσης θα αλλάξει και ο προπολογισμό ε, για να μπορέσει να υλοποιηθεί ό,τι προτείνω. Εν κατακλείδη. Θεωρώ ότι εάν εγκριθεί το Σεπτέμβριο αυτή η γνωμοδότηση, η Επιτροπή μας μπορεί να κλείσει κάποιους συνδεσμούς οι οποίοι ε, θα γίνουν αποδεκτοί από την Επιτροπή των Προϋπολογισμών και από τους ε, εισηγητές του Προϋπολογισμού, ακριβώς όπως έγινε και τα προηγούμενα χρόνια με τις προτάσεις μας. Κατόπιν στην της είναι καθήκον μας τέτοιες προτάσεις να τις ε, προωθούμε για τον προπολογισμό αναλαμβάνουμε επομένω και σε αυτό το μέτωπο τι ευθύνε μα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ, Πίτερ, λέει ο και τώρα πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Κέλλερ, θα ήθελα να πω το εξή. Αρχή-αρχή σα είπα ότι η προθεσμία είναι η 19η Εβδόμου για τι τροπολογίε, ακόμα και αν αλλάξουμε τι ψήφισε. 19 Εβδόμου για τι τροπολογίε. Αυτό δεν αλλάζει, ό,τι άλλο και αν αλλάξει. Κυρία Κέλλερ. Συζητήσαμε το, το αίτημα αυτό της Γενικής Διεύθυνσης για περισσότερους πόρους, οπότε θα είναι πρόβλημα εάν θα, θα, πρέπει να, να τα καταφέρουμε σε όλα αυτά τα μέτωπα, γιατί πώς να γίνουν όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις εάν δεν υπάρχει χρόνος να, για να μελετήσουμε ε, το, το, τα, τα τόσο τεχνικά έγγραφα. Οπότε, για αυτό το πρόβλημα, αυτό το οποίο θα ήθελα είναι να προτείνω ένα πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο ελπίζω θα το υποστηρίξουν οι πολιτικές ομάδες γιατί χρειάζεται να υπάρχει καλύτερη, ε, καλύτερη, καλύτερη παρακολούθηση να μπορούμε να παρακολουθήσουμε καλύτερα τα, τα όσα γίνονται και με τρόπο συστηματικό και χρειάζονται πληροφορίε, ούτω ώστε να έχουμε τι συγκρίσει, να μπορούμε να συγκρίνουμε λοιπόν τα, τα, τις εμπορικέ συμφωνίες, ε, να ξέρουμε τι γίνεται όσον αφορά ε, τα, τα, τα πρότυπα, πώ δικαιολογούνται, ε, όλες τις πτυχές όλων των εμπορικών συμφωνιών και δεν είναι δυνατόν ε, να μας δίνουν τις πληροφορίες οι λομπίστες, η Α, η Β, η κυβερνητική οργάνωση. Πρέπει να έχουμε κάποιο προσέγγιση συστηματική και ίσως ακούσατε για το Finance Watch που συστηματικά παρέχει πληροφορίες όσον αφορά την οικονομική κρίση, τα οικονομικά, τα χρηματοοικονομικά, όλα αυτά που είναι τόσο σημαντικά για την ε, δουλειά μας και δουλειά της Οικονομικής Επιτροπής και οπότε είπαμε ότι όντως μας χρειάζονται τέτοια πράγματα για το ε, για, για, τη δουλειά μας γενικά, για, όλα τα όσα κάνουμε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών είναι διαφορετικός. Δεν, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ε, χρειάζεται και το Trade Watch και ε, ο διάλογος με την κοινωνία των πολιτών ε, οργανώνεται και έτσι μας, μας λέει τι σκέφτεται ο πολίτης και αυτό είναι χρήσιμο για την Κομισιόν αλλά εμείς θα πρέπει να έχουμε αναλυτική γνώση, θα πρέπει να, να ξέρουμε τι γίνεται από κάποιον αμερόληπτο, από κάποιον ανεξάρτητο, αντικειμενικό. Ε, έτσι θα, έχουμε βοήθεια στο έργο μας. Και κατά αυτόν τον τρόπο Νομίζω ότι το σημαντικό είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα του έργου μας, να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε όλες αυτές τις εμπορικές συμφωνίες. Αυτό είχα να σας πω. Κύριε Στάσνη, ίσως ε, κατεβάσω και κάποιες τροπολογίες, αλλά όντως θα χρειαστεί χρήμα για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την αναλυτική υποστήριξη και να κάνει αν όχι πιο εύκολη τη ζωή μας τουλάχιστον θα, θα την κάνει πιο τεκμηριωμένη. Ευχαριστώ. Κύριε Μέρφυ. Ευχαριστώ τον ε, εισηγητή αλλά και με αυτά που είπε η κυρία Κέλλερ ε, συμφωνώ γιατί το Trade Watch θα μας βοηθήσει. Έχω τώρα τρία συγκεκριμένα θέματα για την γνωμοδότηση να σας αναφέρω. Δεν ε, ίσως είναι θέμα διατύπωσης, θέμα γλωσσικό για το σημείο 3. Έτσι όπως τώρα είναι διατυπωμένο το 3, προκύπτει ότι θέλουμε περικοπές στον προπολογισμό. Προσοχή. Προσοχή να αλλάξουμε τη διατύπωση για να μην φαίνεται ότι η διάταξη αριθμών 3 ζητεί περικοπές σε σχέση με εμπόριο και σε σχέση με επίσημη συνεργασία. Τώρα, όσον αφορά την αύξηση της πληκοδότησης για το Aid for Trade, ε, να μην γίνει αύξηση εις βάρος ε, εις βάρος της αναψυχιακής ε, βοήθειας. Το θέμα δεν είναι πόσα χρήματα δίνονται, το θέμα είναι πού πάνε τα χρήματα. Προσοχή, γιατί προωθούν οι μεγάλες εταιρείες νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Εμείς θέλουμε βιώσιμη ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη, οικονομική πολυμορφία, πιο πολλέ θέσει εργασία, αύξηση ιδιωτικού επίπεδου. Αυτά θέλουμε. Και αυτά θα υποστηρίξουμε. Ευχαριστούμε κύριε Μέρφυ. Ποιο τυπώνει. δεν ξέρω εσεί θα μιλήσετε, γιατί έχω εδώ πέρα κατάλογο με τρεις εκπροσώπους κομισιών. Ποιο εξ όλων θα μιλήσει. Εγώ ευχαριστώ, Πρόεδρε, λέει ένας εκπρόσωπο τη Επιτροπή. Εμεί Εμείς λαμβάνουμε υπόψη θα το βλέπατε και ξέρετε και εσείς τις δικές μας θέσεις και γι' αυτό και θεωρούμε ότι εάν υπάρχει τέτοιου είδους ε, συμφωνία για επιπλέον ε, εποπτεία, βεβαίω και ανάλυση μπορεί να γίνει εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς αυτό προς το παρόν αυτό πιστεύουμε. Ο πρόεδρος, σας ευχαριστώ. Πίτερ, θες να δευτερολογήσεις. Στάση. Πάρα πολύ σύντομα, πρόεδρε. Και ευχαριστώ τους συναδέλφους για τα όσα παρατήρησαν, για τα σχολιά τους, για τις προτάσεις τους και όλα, όλα αυτά θα τα εξετάσω από πλευράς των όσων έχουμε εδώ θεωρώ ότι θα πρέπει κάθε πρόγραμμα, κάθε πρόγραμμα να το μελετούμε. Κοιτάξτε, δεν θέλω να ξεφύγω τον προπολογισμό. Αν ζητάμε κάτι για το εμπόριο, είναι ότι ξέρουμε ότι το εμπόριο αποτελεί την προστιθέμενη αξία. Το εμπόριο δίνει θέσει απασχόληση. Το εμπόριο τονίζει την οικονομική ανάπτυξη. Αν κανεί έχει αναπτύξει 2% ρυθμό που πάει στο 3% εάν ε, ε, πάει σε, σωστή, σε άσκηση εμπορικές πολιτικές. Άρα μιλώ τώρα για επένδυση εις των πολιτών. Μερικές φορές θα πρέπει να γίνεται έγκαιρα η επένδυση και να συνεχίζεται μια πορεία και κατά αυτόν τον τρόπο να μπορούμε σε συνεργασία με εταίρους, με γείτονες να προχωρούμε ούτω ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό τον, τον ε, κύκλο της κρίσης τριετή, τετραετή, πενταετή, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με το εμπόριο. Να καταλήξουμε σε κάτι ωφέλιμο, σε κάτι βιώσιμο, όχι μόνο για τους πολίτες, αλλά και για τις χώρες εταίρους. Θα εξετάσω αυτές τις προτάσεις, θα ζυγίσω την καθεμία, ε, τα υπέρ και τα κατά εκάστης. Ο πρόεδρος. Χωρίς μικρόφωνο. Deadline for amendments. 3η Αυγούστου είναι οι πρωτη και 3 Ενάτου θα εγκριθεί το σχέδιο εκθέσεως. Καλώς. Το επόμενο θέμα. 10. Μία στρατηγική ψηφιακή ελευθερία στην εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξέταση του σχεδίου γνωμοδότησης. Τι είναι, ε, επί της ουσίας, ε, ΑΦΕΤ, Αμέλια Άντερς Ντότερ είναι η κυρία, η συγκεντρία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Με αυτή την ευκαιρία να σας παρουσιάσω το σχέδιο κειμένου. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση η οποία έρχεται να συμπληρώσει τα όσα κάνει η ΑΦΕΤ για τη στρατηγική ψηφιακής ελευθερίας. Και εμείς πέραν των όσων κάνει η Επιτροπή Εξωτερικών, θέλουμε να στοχεύσουν περισσότερο στα θέματα εμπορίου. Ασχολούμαστε επομένω με τη ροή των πληροφοριών και λέμε ότι προβληματιζόμαστε. Ανησυχούμε γιατί ακόμα πολυμερός και διμερός συνεχίζουν τη διαμοντεύση με πολλές χώρες. δεν προσέχουμε τα θέματα του copyright. Έτσι βάζουμε φραγμούς στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Την άλλη μεριά, δίνεται στην ε, εφαρμογή της νομοθεσίας Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, έχουμε ανισορροπίες στην εναρμόνιση. Ε, αυτό σημαίνει ότι και οι πολίτες και οι εμπορευόμενοι έχουν πρόβλημα όσον αφορά το copyright και άρα την άσκηση ε, ε, του εμπορίου, την οικονομική δραστηριότητα, αυτά τα οποία επιδιώκουν. Οπότε, γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με αυτές τις εμπορικές συμφωνίες με κάποιες χώρες οι οποίες είναι πάρα πολύ περιοριστικές σε σχέση με ε, ε, τα δικαιώματα τη γιατί υπάρχει κάποια μεγάλη μεγάλη χώρα στην Ανατολή που μπλοκάρει, μπλοκάρει, απαγορεύει την ροή των πληροφοριών μεταξύ πολιτών κλπ. κλπ. Αυτό είναι πρόβλημα για το εμπόριο τη επιχειρήση, αλλά να γίνει προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να εξασφαλίσουμε ότι η δική μας πάροχη δεν θα πρέπει να εμποδίζονται από αυτή τη λογοκρισία. Άλλο θέμα και αυτό. Επίσης, καλούμε να καταρτιστεί μία ατζέντα εμπορική που να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και έτσι να υπάρχει προσβασιμότητα στο διαδίκτυο χωρίς περιορισμούς. Αυτό αφορά τους Ευρωπαίους, αυτό αφορά τις επιχειρήσεις, αλλά φαντάζομαι συμφωνούμε όλοι ότι η ελευθερία της επικοινωνίας και της έκφρασης γνώμης είναι βασικό για την ε, για τη δημοκρατία. Άρα εδώ χρειάζεται κάποια συνέργεια. Τελευταίο τώρα, σημείο αυτής της νομοδότησης αφορά τις εξαγωγές, αφορά ε, τους ελέγχους για τις ε, εταιρείες, μια που οι εταιρείε ε, και εδώ θέλουν να μπορέσουν να προβούν στις κατάλληλες εξαγωγές. Στο δεύτερο σημείο ρώτησε τώρα αναφέρεται κάτι το οποίο είπε η κυρία Νέλη Κρούς. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ακριβές. Λέει ότι το copyright Έχω αρκετή πείραμα για αυτά τα θέματα και αισθάνομαι ότι δεν είναι καλό να παρουσιάζονται στρεβλά οι θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορεί να υπάρχουν κάποια ίσονο σημασία θέματα που μπορούν να αλλάξουν και κάποια άλλα σημεία αν βρούμε καλύτερη διατύπωση για ένα εδάφιο συγκεκριμένο. Αλλά γενικά θα έλεγα ότι είναι ενδεικτικό αυτό και εκπροσωπεί το πώς βλέπουμε τα θέματα του ευρωπαϊκού εμπορίου, πώς θα έπρεπε να στοχεύουν και να διαμορφώνονται αυτά. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ, Κρίστοφερ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Σκιώδης συζητητής από το ΕΛΚ. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποια σχόλια. Λοιπόν, πιστεύω ότι είναι ένα τεράστια σημασία ε, ζήτημα αυτό και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα μπορούσε κανεί να τοποθετηθεί και να αναπτύξει τα θέματα τη ψηφιακή ελευθερία επί ώρε. Βλέπω κουνάει το κεφάλι του ο πρόεδρο. Δεν το κάνω, δεν μιλήσω επί ώρε. Είναι όμω σημαντικό για τα μέλη αυτή τη κοινοβουλευτική επιτροπή να αποσαφινιστεί ότι ένα ανοιχτό θέμα στο διαδίκτυο έχει, θέμα, έχει σπουδαιότητα για το εμπόριο γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος της οικονομίας διεξάγεται στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στο διαδίκτυο, online και περιορισμοί σε σχέση με αυτή την πτυχή περιορίζουν το εμπόριο. Υπάρχουν και θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχουμε και ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή που σίγουρα θα τονίσει την πτυχή των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Είναι η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Είναι όμως το θέμα να δούμε τι θα κάνουμε με τις δικές μας αρμοδιότητες για το εμπόριο ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Η διάσταση για το εμπόριο, η συνιστόσα στο εμπόριο, το να περιορίζει κανείς το διαδίκτυο, περιορίζει το ε, εμπόριο. Τώρα, η ε, τα τείχη τα οποία υψώνονται για να προστατευθούν κάποιοι, ε, ε, βλέπουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για προστατευτισμό, για προστα... χρήση για στρεβλό προστατευτισμό. Η Κινέζικη κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν αυτό το μέσο επικαλούμενες λόγους ε, εθνικής ασφάλειας και άλλα τέτοια προσχήματα. Όμως ο κύριος στόχος είναι να υπάρξει προστατευτισμός, να δημιουργήσουν τύχη ώστε να προστατεύουν τα δικά τους συμφέροντα και τα δικά τους μέσα στο εμπόριο και να περιορίζουν την πρόσβαση σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις στο εμπόριό τους. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που πραγματικά αυτή η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή πρέπει να λάβει υπόψη. Το θλιβερό είναι το ότι αυτή η ε, γνωμοδότηση χάνει αυτή τη συνιστόσα από το θέμα ουσίας. Δηλαδή απουσιάζει το θέμα του ψηφιακού προστατευτισμού που ο ψηφιακός προστατευτισμός είναι ένα μεγάλο εμπόδιο στην ευρωπαϊκή οικονομία. Δίνεται μεγάλη έμφαση στα θέματα της ε, ε, ψηφιακής ε, των προσωπικών πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων ως θέμα που μπορεί να περιορίζει την ψηφιακή ελευθερία. Η ελευθερία πρέπει να είναι σεβαστή όμως όταν βλέπουμε ότι υπάρχουν εξορισμού κάποια εμπόδια για την ελευθερία πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Περιοριζόμενος τώρα στα θέματα της πτυχής των δικαιωμάτων του ανθρώπου σε σχέση με περιορισμούς στο διαδίκτυο. Κάνοντας λόγο για τη Λευκορωσία ή σε σχέση με τους εκπροσώπους της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την ε, Λευκορωσία, δεν είναι μόνο τα θέματα των ε, προσωπικών πληροφοριών ή θεμελιωδών δικαιωμάτων, το θέμα του κλεισίματος ε, των περιορισμών που υφίστανται. Είναι ο περιορισμός στο Facebook της πρόσβασης στο facebook και άλλες δυνατότητες ε, περιαγωγής και αναζήτησης στο διαδίκτυο που πάλι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για τον προστατευτισμό. Έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη ε, για το e-site από ειδικά οργανισμό που λέει ότι μπορεί να προσφύγει κανείς στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για τέτοιου είδους περιορισμού. Μια και, το, μια και έχει αποτελεσματικά μέσα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου για να πιέσει για ανοίγματα και πολλές από αυτές τις χώρες έχουν αναλάβει δεσμεύσεις όσον αφορά τα πνευματικά δικαιώματα και τις, ε, τα δικαιώματα παραγωγών, γκάτς, πνευματικής ιδιοκτησίας Δύο παρατηρήσεις θα ήθελα να κάνω επιπλέον. Πρώτον, πιστεύω ότι υπάρχει ένα ουσιώδες στοιχείο ότι όσον αφορά το εμπόριο και τον εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών, πολλά πράγματα είναι αντικείμενα μιας χρήσης, μονής, όχι διτής χρήσης. Και Πολλά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σε αυτό το πλαίσιο. Αν όμω μια υπηρεσία πάροχος τηλεπικοινωνιών παρέχει υπηρεσίες στη Λευκορωσία, για παράδειγμα, έχουν ηθική τουλάχιστον υποχρέωση για να προβληματιστούν και να δουν πώς αυτές οι υπηρεσίες θα αντιμετωπίζονται από τις κυβερνητικές αρχές, από την κυβέρνηση δεν θα ήταν προς ικανοποίηση κανενός ε, αν δεν ε, μπορούσε να προαχθεί η ελευθερία ε, της χρήσης με τη χρήση τέτοιων εξοπλισμών εκεί. Θα έπρεπε όμως να επιτηρεί κανείς και να εποπτεύει το εμπόριο με τέτοιες χώρες όσον αφορά τις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχονται. Υπάρχει εδώ ένα θέμα ουσίας Ίσως θα μπορούσα να το διατυπώσω διαφορετικά, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Εν πάση περιπτώσει δεν με την άποψη ότι δεν θα έπρεπε να συνάψουμε εμπορικές συμφωνίες που να συνάπτονται με το IGR ή με άλλα ψηφιακά κεφάλαια προτού υπάρξει ένα είδους συνένεση στην Ευρώπη για όλα αυτά τα θέματα. Θα ήταν πάλι ένα πρόσχημα να πει κανείς δεν μπορούμε να έχουμε μια σφαιρική συμφωνία. Παράδειγμα, για τις κλιματικές αλλαγές, προτού έχουμε ευρωπαϊκή συνένεση πώς θα αντιμετωπιστούν τα θέματα των κλιματικών αλλαγών. Ε, τότε δεν θα υπάρξει ποτέ συνένεση πώς ακριβώς θα πρέπει να αντιμετωπιστούν οι κλιματικές αλλαγές. Και ποτέ δεν θα μπορέσουν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό όλες οι συμφωνίες πρέπει να βασίζονται στο κεκτημένο στο κοινοτικό και εκτιμένο. Αυτό που κάνουμε σήμερα με τον Καναδά για τις συμφωνίες εμπορίου σήμερα βασίζεται στο κοινοτικό και εκτιμένο και έτσι θα πρέπει να διαπραγματευόμαστε και να ολοκληρώνουμε τις διαπραγματεύσεις και τις συμφωνίες με βάση το, το κοινοτικό και εκτιμένο. Έτσι πρέπει να προχωράμε και στους πιο σημαντικούς τομείς που είναι οι υπηρεσίες, η παροχή υπηρεσιών στον ψηφιακό τομέα. Θα ήταν αντιπαραγωγικό και θα αντέβαινε το ευρωπαϊκό συμφέρον αν κάναμε κάτι διαφορετικό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Κρίστοφερ. Η κυρία Μπαντία Κουτσέ, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η έκθεση για τη στρατηγική για την ε, ψηφιακή ελευθερία στην εξωτερική πολιτική είναι πάρα πολύ σημαντική σήμερα και πιο συγκεκριμένα μετά από την απόρριψη της ΑΚΤΑ στο Στρασβούργο την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι πολύ καλές οι θέσεις της εισηγήτριας που υποβάλλονται στην ίντα και ορίζονται οι προτεραιότητες για την ψηφιακή ελευθερία. Θέλω όμως να επιμείνω σε κάτι ότι ο, τερινός, ο τωρινός κατακαιρματισμός της στρατηγικής ε, για τα πνευματικά δικαιώματα πρέπει να διορθωθεί και πρέπει να ορίσουμε ένα σύστημα κοινής προστασίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτό το θέμα δεν βρίσκεται μέσα στην έκθεση αλλά συνδέεται με την έκθεση και με αυτή τη στρατηγική. Θα πρέπει επίσης να αυξήσουμε την περιφρούρηση για την οσιρότητα της τεχνολογίας που μπορεί να προέρχεται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, δεσμεύσεις που έχουμε στα διεθνή φόρα Επίσης, το ρόλο που μπορεί να παίξει η Ένωση για την ψηφιακή ελευθερία σε κοντινές χώρες και σε τρίτες χώρες με τις οποίες έχει συνάψει εμπορικές συμφωνίες. Πιστεύω ότι η ελεύθερη κυκλοφορία κατάρτισης και εγκατάστασης είναι ουσιαστική στο πλαίσιο των εμπορικών ανταλλαγών. Αυτές είναι οι ιδέες που θέλω να θέσω και συγχαίρω την εισηγήτρια γιατί έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά και επίσης την ευχαριστώ για τη συνεργασία της. Κανείς από τους φιλελεύθερους το ECR στη συνέχεια για την ανάγνωση των παρατηρήσεων αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος ε, το διαδίκτυο της καθημερινής ζωής. Οι προκλήσει όμω του ψηφιακού κόσμου που σας αποκαλούμε σε διευρυμένο πλαίσιο αποτελούν εν δυνάμει κατά τα τελευταία 5-10 έτη ένα μεγάλο πλαίσιο. Είναι ένα ε, νέο παρθένο έδαφος ε, το διαδίκτυο. Καλούμαστε λοιπόν να αποφασίσουμε πώς θα μπορέσει να ρυθμιστεί και σε πολλές περιπτώσεις αν κάποια μορφή ελέγχου ή όχι χρειάζεται και πώς θα πρέπει να λειτουργήσει. Όταν έχουμε το θέμα δημιουργίας ευημερία και πλούτου για όλους θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το ψηφιακό θεματολόγιο της Ευρώπης ψηφιακή ημερήσια διάταξη και οι θετικές επιπτώσεις ε, που μπορεί να έχει, να χρησιμοποιείται υπέρ της δημιουργικότητας και καινοτομίας για να παρέχει οικονομική ανάπτυξη υψηλής προδιαγραφής, ε, υψηλών προδιαγραφών και ποιότητας αναβαθμισμένες θέσεις ε, εργασίας κτλ. Ωστόσο για την, το ψηφιακό θεματολόγιο στην Ευρώπη πρέπει να έχουμε ισόρροπες σχέσεις μεταξύ IPR και των συμφερόντων των πολιτών για την προσπελασιμότητα, την πρόσβαση σε θέματα θέματα ουσίας και γνώσης. Όταν έχουμε το θέμα διαπραγμάτευσης για διεθνείς συμφωνίες, οι επιχειρήσεις μας που παράγουν αγαθά οι υπηρεσίες θα πρέπει μέσω αυτού του τρόπου του, του IPR να μπορούν να προσαρμόζονται σε, στις ανάγκες και τα πρότυπα. Υπάρχει ένα επιχείρημα ότι σε ένα κόσμο όλο και μεγαλύτερης επεξεργασίας λεπτομεριών, η αύξηση αποθήκευσης όσον αφορά ε, ψηφιακά τέτοια προϊόντα πολλές φορές ε, δεν προσεγγίζει παρά ένα πολύ χαμηλό επίπεδο. Θα πρέπει ως νομοθέτες να επιτρέπουμε τους παρόχους ε, τέτοιων υπηρεσιών ουσίας να μπορούν να παρέχουν σε, με αναλογικότητα τα προϊόντα τους, όμως να μην δώσουμε την δυνατότητα κάποιοι να ε, εκμεταλλεύονται με στρεβλό τρόπο τις δυνατότητες. Θα πρέπει τα πρότυπα, τα επιχειρησιακά να συνεπάρχουν και θα πρέπει η αγορά να αποφασίσει ποιο θα επικρατήσει και ποιο θα επιλέγεται. Αυτά από πλευράς του Σαϊτ Καμάλ. Ο κύριος Χέρμουτ Σόλτς παρακαλώ έχει τον λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να καλωσορίσω για αυτή την ε, έκθεση γιατί μετά από τη φάση από την οποία περάσαμε μετά από τη συμφωνία ΑΚΤΑ έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η γνωμοδότηση και σε σχέση και με την ε, ΑΦΕΤ θα ήθελα να ενημερώσω ότι έχουμε ήδη μια διεργασία που ξεκίνησε από τον εισηγητή της ΑΦΕΤ και που είναι αναπληρωματικό μέλος επίσης και στη δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή ο Ευρωβουλευτής όλοι οι εισηγητές και σκιώδεις εισηγητές και Όλοι όσοι ενδιαφέρονται και εμπλέκονται από πλευρά άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών προσκαλούνται να συμμετάσχουν για να συζητήσουν και να δημιουργήσουν μια κοινή πλατφόρμα για την εξέταση αυτού του ευρύτερου θέματος. Διότι είναι σωστό ότι πρέπει να συμμετάσχουμε και ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου μέσα σε αυτά τα πλαίσια και τα θέματα τα οποία αναφέρονται και θίγονται εδώ και από πλευράς ε, των παρεμβάσεων έχουν ιδιαίτερη εμβέλεια, έχουν μεγάλο εύρος και αν και όταν ο κύριος Φιέρνερ αναφέρεται στα θέματα των δικαιωμάτων των πολιτών και δικαιωμάτων του ανθρώπου, θέλω να υπενθυμίσω ότι προέρχομαι αρχικά από μια χώρα που βρισκόταν υπό το μποϊκότ του καταλόγου COCOM για το Ανατολικό Μπλοκ, όπου τεχνολογία των υπολογιστών και άλλα τέτοια θέματα δεν επιτρεπόντουσαν να προάγονται σε σχέση με τις χώρες μας. Ξέρω από την κοινωνία και την προηγούμενη χώρα στην οποία ζούσα τι σημαίνουν αυτά τα πράγματα. Αν λέμε ότι δεν πρέπει μόνο οι αγορές να αποφασίζουν, αλλά πρέπει να ρυθμίζονται αυτά τα πράγματα από ρυθμιστικούς μηχανισμούς και διατάξεις, πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και συνετοί. Για αυτή τη γνωμοδότηση θέλω να υπογραμμίσω, πιστεύω, το θέμα 3, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να παραμείνουμε εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το πλαίσιο. Να βρούμε μια προσέγγιση, να αποσαφηνίσουμε τα πράγματα όπως πρέπει. Ιδιαίτερα μετά από αυτά που συνέβησαν με την Άκτα και τα μαθήματα τα οποία αναγκαστήκαμε να συναγάγουμε από αυτή τη διαδικασία της Άκτα, της συμφωνίας αυτής. Πρέπει στα πλαίσια διεθνών συμφωνιών να βασιζόμαστε στις εσωτερικές μας προσεγγίσεις και την εσωτερική συνένεση και συμφωνία που υπάρχει στο Ευρωκοινοβούλιο, στο Δικαστήριο, στα κράτη-μέλη, από τους πολίτες μας. Δηλαδή αυτό πιστεύω ότι πρέπει να είναι πραγματικά πολύ σημαντικό στοιχείο. Δεύτερον, θα ήθελα να πω, να προτείνω κάτι, να παραμείνουμε στο διεθνές πλαίσιο στο οποίο πρέπει να αναπτύξουμε αυτό το θεματολόγιο, αυτή την ημερήσια διάταξη. Υπάρχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου, υπάρχει το Διεθνές Γραφείο Εργασίας. Αυτά θα πρέπει να αναφέρονται στο, στη γνωμοδότησή μας. Και υπάρχει επίσης και το θέμα των ψηφιακών ελευθεριών στην εξωτερική πολιτική. Και αυτό θέτει ζητήματα, εδώ συχνά συζητάμε για την αναπτυξιακή βοήθεια, για την ανάπτυξη όταν κάνει κανείς λόγο για το διεθνές εμπόριο, πάντα έχουμε το πρόβλημα ότι έχουμε ιδιωτικό τομέα ιδιωτικής χρήσης δηλαδή και την ιδιωτική ιδιοκτησία, η κυριότητα σε κάποια μέσα για την παροχή υπηρεσιών στο διαδίκτυο παρόχους που βρίσκονται υπό ιδιωτική ιδιοκτησία και κυριότητα και για την διάχυση και ανταλλαγή πληροφοριών, στοιχείων, ενημέρωσης, γνώσης, πρέπει να βρούμε ένα ισορροπημένο τρόπο αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις αυτές να διασφαλίσουμε από πλευράς νομοθέτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση πώς θα πρέπει να ρυθμίζονται αυτά τα θέματα. Είμαι πρόθυμος να το κάνουμε αυτό και με ιδιαίτερη ικανοποίηση να συνεργαστώ με τον εισηγητή να έχουμε μια καλή γνωμοδότηση από την Επιτροπή μας τελικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σε τρία σημεία παρατηρήσεις. Πρώτο, πραγματικά η ελευθερία στο διαδίκτυο είναι μια ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη, αλλά επίσης και για τη συμμετοχή και με ένα, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Αλλά δεν συμβαίνει αυτόματα αυτό. Έχουμε στην Ευρώπη σίγουρα λύσεις για ένα ασφαλές ε, εμπόριο στο διαδίκτυο, ηλεκτρονικό εμπόριο. Αλλά έχουμε και λύσεις για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών, των εμπλεκομένων στο διαδίκτυο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Και αυτό πρέπει και παγκόσμια να προαχθεί. υποστήριξη λύσεων hardware και software που θα διασφαλίζουν ασφαλές ε, ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικό διεθνές εμπόριο και θα διασφαλίζει την συμμετοχή των ανθρώπων, των πολιτών σε αυτές τις διεργασίες. Και υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες τέτοιες τεχνικές λύσεις. Σε κάποια κρατήδια στην Γερμανία και κάποιες περιφέρειες το κάνουμε αυτό. Ζητείτε οι άνθρωποι να ψηφίζουν μέσω διαδικτύου και να επιλέγουν ποιες διαδικασίες ε, προτιμούν. Και κάτι τέτοιο θα πρέπει και προς τα έξω να προαχθεί από εμάς με ιδιαίτερο τρόπο. Δεύτερη παρατήρηση κύριε Φέρνερ. Ελπίζω ότι σας κατάλαβα καλά σε αυτό που είπατε. Το σημείο 6 την χάνει υποστήριξη από πλευρά σας. Ότι εφ' εξής, στη συνέχεια μια εξέταση Εξάντε θα πρέπει να γίνεται, εκ προημίου δηλαδή, για ψηφιακό εξοπλισμό και τέτοιου είδους τεχνολογίες, ακριβώς για χώρες όπου υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τη χρήση και εκμετάλλευση αυτών των εξοπλισμών και συσκευών. Ήδη έχουμε συζητήσει μία φορά για το θέμα για την έκθεση διπλής χρήσης, διτής χρήσης. Δυστυχώς δεν υπήρξε εκεί η πλειοψηφία για μία εξέταση εξ εκ προημίου παρότι στην αναθεώρηση του κανονισμού διτής χρήσης κανονικά θα πρέπει κανείς, θέτει κανείς το αίτημα μιας τέτοιας εξέτασης και ελπίζω ότι από κοινού μπορούμε να εγκρίνουμε αυτή την αρχή για να είναι σαφές ότι δεν θέλουμε να έχουμε περιορισμού στις εξαγωγές και δεν μπορούμε εμείς να αποφασίζουμε ποια συσκευή και ποιος εξοπλισμός θα χρησιμοποιείται για, για ποια χρήση αλλά σε κάποιες χώρες πρέπει προτού δώσουμε άδεια εξαγωγής τέτοιων προϊόντων να εξετάζουμε πιο πριν αν πρέπει να δοθεί μια τέτοια άδεια ή όχι δεδομένων των συνθήκων και προϋποθέσεων. Τρίτο, το θέμα της προστασίας ε, πνευματικών δικαιωμάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή πνευματικής ιδιοκτησίας αν δεν υπάρχει λύση να μην προχωράμε δεν οδηγεί πουθενά, διότι επί 20 χρόνια μπορεί να συνεχίζεται μια τέτοια τροχοπέδηση, ένα τέτοιο πρόβλημα. Πρέπει να κληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιο έντονα από εμά, το δυνατόν γοργότερα να ε, προστατεύσει με πιο αποτελεσματικό τρόπο τα πνευματικά δικαιώματα ιδιοκτησία στον ψηφιακό τομέα. Άκουσα από το μίση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο Επίτροπο Μπαρνιέ λέει σε αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο τη αρμοδιότητα τη Επιτροπή δεν προτίθεται να το κάνει αυτό. Έχει φόβο, φοβάται το ίδιο του το θάρρος και δηλιάζει να υποβάλει μια τέτοια πρόταση και να την προαγάγει. Πρέπει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακριβώς σε σχέση με τις διεθνείς συμφωνίες να ζητήσουμε να εμπλακεί πιο έντονα και να ζητήσουμε πιο γοργά να υποβληθεί μια πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διασφάλιση πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων παραγωγών και δημιουργών στο διαδίκτυο. Μπορεί ίσως να μας ενημερώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν ο ψήθυρος η φήμη αυτή ότι σε αυτή την κοινοβουλευτική θητεία δεν θα υποβάλει πρόταση ο κύριος Μπαρνιέ σχετικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μπέρντο. Κρίστοφερ. Δεν νομίζω ότι διαφωνούμε και θέλω να το πω αυτό. Μπορεί για τη διτή χρήση να είχαμε, αλλά όχι σε αυτόν τον τομέα υποχρεωτικά. Διότι η πρόκληση που βλέπω σε αυτόν τον τομέα δεν είναι το θέμα της χρήσης, ε, διτής χρήσης αυτών των συσκευών και εξοπλισμών. Παράδειγμα, είχα πολλές συζητήσεις ε, με την Ericsson που παράγει εξοπλισμό στον ε, ε, διακοπτών και άλλων, άλλου εξοπλισμού στις τηλεπικοινωνίες οι νέες δυνατότητες καθιστούν εφικτό για τις νομικές αρχές επιβολής του νόμου ε, σε όλες, μια και σε όλες τις χώρες στην Ευρώπη οι κυβερνήσεις επιτρέπεται υπό κάποιους όρους και συνθήκες να παρακολουθούν συνδιαλέξεις τηλεφωνικές και να παρακολουθούν ε, τα όσα γίνονται. Αυτό είναι κάτι το δεδομένο σε σχέση με αυτούς τους εξοπλισμούς. Το πρόβλημα όμως είναι αν πουλήσουμε αυτούς τους εξοπλισμούς σε κάποιες ε, χώρες που δημιουργούνται προβλήματα. Το, για παράδειγμα στην Λευκορωσία που είχαμε και τη συζήτηση με την ε, Τελεσόνερα που έχουν τέτοιου είδους υπηρεσίες ε, στη Λευκορωσία να επιτρέπεται τώρα η μυστική υπηρεσία να εγκαθίσταται στην έδρα ή στο, στην θέση αυτή και να παρακολουθεί τις συνδιαλέξεις και τα τεκτενόμενα έχει δίκιο ο Χέιμουρ Σόλτς που λέει το να μην πουλάμε τέτοιου είδους εξοπλισμό ή ε, συσκευές ή να μην λειτουργούμε σε τέτοιες χώρες θα το καθιστούσε ακόμα δυσκολότερο για τις δυνάμεις που θέλουμε να υποστηρίξουμε, διότι οι δημοκρατικές δυνάμεις χρειάζονται το διαδίκτυο και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Είναι λοιπόν θέμα ισορροπιών εδώ που πρέπει να αναζητηθούν και δεν μπορούμε ισοπεδωτικά να δράσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε «Α, αυτό να μπει στο παράρτημα των ε, αντικειμένων για τη διτή χρήση». Πρέπει να διεξαχθεί μια συζήτηση να δούμε πώς θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε επί τόπου. Αλλά ταυτόχρονα να γνωρίζουμε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτι τέτοιο στρεβλά. Εν πάση περιπτώσει, είναι ένα τεράστιο ζήτημα αυτό το IPR και θα μπορούσαμε επί ώρες να το συζητούμε. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν νομίζω ότι αυτό είναι το μείζον θέμα όσον αφορά τις ψηφιακές ελευθερίες ε, στο διαδίκτυο και στις εμπορικές σχέσεις. Και θα έλεγα ότι η ιδέα του να υπάρξει συνένεση Πιστεύω ότι χρειάζεται μια μεταρρύθμιση IPR. Χρειαζόμαστε μια δυναμική αλλαγών και μεταβολών στο IPR διότι οι οικονομικές αλλαγές και μεταβολές, η κατανάλωση αυτών των ζήτηση και κατανάλωση αυτών των αγαθών, σε δέκα χρόνια θα έχουν αλλάξει όλα αυτά τα πλαίσια. Δεν θα ισχύουν αυτά που ισχύουν σήμερα. Το να πιστεύει κανείς ότι θα μπορέσει να εξευρεθεί μια συνένεση και μετά θα είναι εσαΐ δυνατό να προχωρήσουμε και να ασχοληθούμε με τα θέματα εμπορίου είναι κάπως αφελές θα έλεγα, σίγουρα αφελές θα έπρεπε όλες οι διαπραγματεύσεις πάντα να βασίζονται στο κεκτημένο και μετά να προσαρμόζεται και να αλλάζει αυτό το κεκτημένο, να ξεκινούν μετά νέες διαπραγματεύσεις. Αλλά χρειαζόμαστε συμφωνία από αυτών των σημείων σίγουρα πιο πριν. Ευχαριστώ. Mm. θα ήθελα ένα θέμα να αναφέρω που πιστεύω ότι στη συζήτηση μπορεί να αμεληθεί ίσως και απειλείται να αγνοηθεί Πιστεύω ότι οι συγητές στην παρουσίαση των κεντρικών σημείων επικεντρώθηκαν στο θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας και πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό. Αυτό που εμάς ως ΕΛΚ μας ενδιαφέρει είναι ο τίτλος αυτής της γνωμοδότησης πραγματικά να είναι διαφορετικός. Και ο τίτλος και της πρωτοβουλίας στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που είναι διαφορετικός. Δηλαδή εδώ περί τίνος πρόκειται για μια ψηφιακή ελευθερία στη στρατηγική, στην πολιτική εξωτερικού εμπορίου. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις ελευθερίες ώστε η δημοκρατία, τα δικαιώματα του ανθρώπου, όλα αυτά να προαχθούν στο εξωτερικό μέσω του, των υπηρεσιών αυτών. Μέσω σύγχρονης τεχνολογίας μπορεί κανείς να περιορίσει τις ελευθερίες στο διαδίκτυο, σίγουρα. Αν δει κανεί την κατάσταση στο Ιράν, ότι μαθαίνουμε κάποια πράγματα από το Ιράν παρόλα αυτά, φυσικά χρησιμοποιεί τι δυνατότητε που τεχνολογικά υπάρχουν η κυβέρνηση ώστε να καταπιέσει όσου εμπλέκονται στο διαδίκτυο. Αλλά αν δεν υπήρχε κάποια τέτοια τεχνολογία, κανεί δεν θα μπορούσε να μα δώσει πληροφορίε. Να προβληματιστούμε λοιπόν πώ μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την ψηφιακή τεχνολογία ώστε η διάχυση πληροφοριών, η δημοκρατία, η ανταλλαγή απόψεων να μπορούν να προαχθούν Αυτέ Αυτές οι πτυχέ πρέπει να τύχουν προσοχή και να βρεθούν στο επίκεντρο. Γιατί διαφορετικά κάθε, τεχνική, κάθε τεχνολογία μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο κατάχρηση. Ε, τότε δεν θα πρέπει να εξάγουμε τίποτα στο Ιράν. Κανενό είδου τεχνολογικό προϊόν. Διότι τότε θα έλεγε κανεί ότι είναι αφόρητο το τι κάνουν τα καθεστώτα αυτά. Ε, δεν θα υπήρχαν τότε διάβλοι επικοινωνία. Και δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να έχουμε πληροφορίε και να προχωρήσουμε ε, σε σχέση με τα θέματα αυτό. Για το θέμα εξ πώς τα ή εξ δηλαδή εκ των υστέρων ή εκ, των, εκ προημίου ε, εξέτασης και αδειοδότηση, παρακαλώ να προβληματιστούμε. Μήπω υπάρχει παρανόηση εδώ. Πρώτον, μια, ένας καλός έλεγχος εξ άντε, εκ προημίου, των προηγουμένων. Και υπάρχει λοιπόν αυτή η πτυχή που, είναι, που μπορεί να θέσει θετικές προοπτικές, αλλά μία εκ των υστέρων διεργασία ελέγχου μπορεί υπό κάποιες πτυχές και προϋποθέσεις να είναι καλύτερη. Ας συγκρίνουμε και ας δούμε τι γίνεται σε σχέση με τις εξαγωγές, ε, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, εξπόστα έλεγχος, εκ των υστέρων έλεγχος και εδώ ίσως υπάρχει κάποια παρανόηση για κάποιους. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν εξάγεται και μετά θα πούμε «Α, τι εξάγεται έχουμε εδώ εξαγάγει, κατά λάθο ήταν μια ατομική βόμβα και δεν έπρεπε να είχε εξαχθεί. Αυτό σημαίνει εξ post έλεγχος, εκ των υστέρων έλεγχος, σημαίνει κάποιες επιχειρήσεις, κάποιοι πάροχοι που ξέρουν καλά τους κανόνες και είναι αξιόπιστοι, που επί χρόνια έχει αποδειχθεί τι επιτρέπεται να εξάγουν και τι όχι και το γνωρίζουν αυτό, μπορούν να εμπιστευθούν να ακολουθήσουν τις εξαγωγικές διαδικασίες όπως το έκαναν και εκ των υστέρων να μας γνωστοποιήσουν, μια και είναι νόμιμη αυτή η εξαγωγή, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ανταλλακτικά, εξαγωγές ανταλλακτικών, Πώς μπορούν όλα αυτά στον πρακτικό τομέα να λειτουργήσουν διαφορετικά όταν πρόκειται για ώρες που χρειάζονται να φτάσει ακριβώς την ώρα του το προϊόν, να φτάσει ένα αεροπλάνο ακριβώς την ώρα ή κάποιο προϊόν να είναι τη στιγμή εκείνη διαθέσιμο όπως απαιτείται. Όταν έχουμε αδειοδότηση που έχει ήδη δοθεί και τα λοιπά, όταν απαιτείται εκ προημίου κάτι τέτοιο και μετά από μερικές εβδομάδες δίνεται η άδεια και έχουμε καθυστέρηση, ε, να το λάβουν υπόψη αυτό οι συνάδελφοι στη συζήτηση για τη διτή χρήση και τη συζήτηση που θα διεξαχθεί ούτως ή άλλως για αυτό το θέμα, να προβληματιστούμε και να δούμε το θέμα εξπόστη εξάντε που πριν από 1,5 χρόνο, χρόνο το συζητήσαμε ούτως ή άλλως, αν πρέπει πρέπει να ξανανοίξει ή όχι και τι θα κάνουμε με αυτή τη γνωμοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χέλμουτ θέλεις να επανέλθεις με τις παρατηρήσεις σου. Ναι πρόεδρε. Θα ήθελα μόνο μία πτυχή να αποσαφηνίσω, να διευκρινίσω, διότι κάποια παρανόηση δημιουργήθηκε με αυτή την πτυχή. Αν δούμε τον αγγλικό τίτλο της γνωμοδότησης για αυτή την έκθεση, στην ΑΦΕΤ, εδώ τι βλέπουμε. Έχουμε διαφορετικό τίτλο από τη γερμανική μετάφραση. Δεν πρόκειται αγαπητέ Κασπάρη για τις ε, ψηφιακές ελευθερίες. Πρόκειται για τη στρατηγική για τις, ε, ελευθερίες, για τις ψηφιακές ελευθερίες και ο εισηγητή τη ΑΦΕ την προηγούμενη εβδομάδα στο Στρασβούργο το κατέστησε σαφέ. Περί τίνο πρόκειται. Πρόκειται για δικαιώματα πνευματική ιδιοκτησία, δικαιωμάτων των δημιουργών, των παραγωγών, όλα αυτά τα θέματα που αφορούν το εξωτερικό πεδίο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η αφετηρία, αν τα κατάλαβα σωστά. Και από πλευρά των παρατηρήσεων όσον αφορά την ε, θέση ε, τη εισήγηση ε, τη Επιτροπή Εξωτερικών, σε αυτό επικεντρώνεται. Εμεί εδώ έχουμε τα θέματα εμπορίου στα οποία επικεντρωνόμαστε. Δεν μπορούμε στη γνωμοδότηση για την Επιτροπή Ανάπτυξης ε, να λέμε ότι το εμπόριο πρέπει να καθορίζει τη δική της γνωμοδότηση της Επιτροπής ε, Ανάπτυξης. Πρέπει να επικεντρωνόμαστε σε εκείνα τα θέματα που αφορούν το εμπόριο και τις εμπορικές συναλλαγές να επικεντρωνόμαστε και να δούμε τη σημασία που έχει για αυτά τα θέματα η στρατηγική για την ψηφιακή ελευθερία. Για τέτοια θέματα δηλαδή πνευματικής ιδιοκτησίας και ούτω καθεξής και τα λοιπά. Και με αυτά να ασχοληθούμε. Αυτή είναι η σωστή προσέγγιση που από κοινού με τους εισηγητές για αυτή τη γνωμοδότηση θέλουμε να ακολουθήσουμε και να αναπτύξουμε. thank you, Helmut. I have to say... Ευχαριστώ είναι ένα θέμα που είναι πραγματικά πολύ θελκτικό και ελκυστικό. Μεγάλη συζήτηση, μεγάλου εύρους διεξάγεται. Η Επιτροπή παρακαλώ. No apologies, you will have to bear with me, uh, Mr. Chairman. My name is from uh, DG Trade. Προέρχομαι από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να σας πω ότι συμφωνούμε με τους ε, γενικότερους στόχους του εισηγητή, δηλαδή να εξασφαλιστεί η ελευθερία του λόγου, η ελεύθερη διακίνηση, ε, τη συζητήτρια για το διαδίκτυο όλα αυτά και όπως ο κ. Λάγκε επίσης ε, και από βάση οικονομικής είναι σημαντική η ελευθερία στο διαδίκτυο είναι μια προϋπόθεση επιτυχίας ε, τη σημερινή μέρα είναι ένας από τους στόχους που προσπαθούμε να πετύχουμε με τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου να διευκολύνουμε το εμπόριο Άρα, γι' αυτό σας λέω ότι ε, μας προκαλεί κάπως έκπληξη ε, η μνήμα του να παγώσουν κάποιες ε, διαπραγματεύσεις συμφωνιών. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ποια είναι τα θέματα, για ποιους λόγους προτείνεται αυτό. Γιατί έχουμε τώρα κάποιες διαπραγματεύσεις για το νέο κεκτημένο, το ηλεκτρονικό εμπόριο, τη σχετική οδηγία. Βεβαίως και υπάρχει εγγύησης ελεύθερη χρήση του διαδικτύου για όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και παραπέμπω τώρα στην συμφωνία με την Κορέα. Ισχύει εδώ και ένα χρόνο και από γνωρίζω. Δεν έχει επηρεαστεί καθόλου η ελευθερία του ίντερνετ ε, δεν, δεν έχουμε στοιχεία ότι η Κορέα περιορίζει τη χρήση του Ιντερνετ. Εάν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, να τα εξετάσουμε. Επίσης, ε, αυτό πέτυχε τον κύριο Μπαρνιέ, ε, αυτό αφορά τον κύριο Μπαρνιέ και την Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς. ξέρω εγώ αυτό που ξέρετε και εσείς, τον κύριο Μπαρνιέ δήλωσε ότι θα εξετάσει αυτά τα θέματα, τα θέματα πνευματικής ιδιοκτησία και σε σχέση με το διαδίκτυο θα το κάνει αυτό κατά την τρέχουσα θητεία. Δεν έχω τίποτα άλλο να σας αναφέρω προς το παρόν. Ευχαριστώ. Εισηγήτρια. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τα όσα είπανε, για την ε, ανάλυση που έγινε. Όπως είπατε Πρόεδρε, είναι συναρπαστικό, μεγάλο θέμα, ενδιαφέρον. Νομίζω το καλύψαμε το θέμα πλήρω. Και το υπαριθμόν 6 ε, ε, την ε, χρήση αυτήν, την μοναδική ε, είπαμε ότι ε, έχει χιόρι αυτή η ανάλυση κατά κάποιο τρόπο γιατί πάντως το θέμα είναι πάρα πολύ διφορούμενο ιδίω τώρα, τώρα που έχει απορρίψει το Κοινοβούλιο την συμφωνία για, τα, για την, την άκτα όσον αφορά την, ε, τις απομιμήσεις. Όχι, δεν λέμε ότι πρέπει να σταματήσουν όλες οι για συμφωνίες ελευθερών εμπορίου. Θα πρέπει να είναι αμοιβαία ωφέλιμες, δηλαδή να ωφελούν όχι μόνο την άλλη πλευρά, να ωφελούν και εμάς. Γι' αυτό κάνουμε διαπραγματεύσει, για να ωφεληθούμε και εμεί. Όταν έχουμε τέτοια κατάθμιση στην εσωτερική αγορά, τότε τέτοιε συμφωνίε δεν μα ωφελούν. Νομίζω ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε ε, και ιδίω όταν λέμε στην Κομισιόν και χαράζουμε στην νέα πολιτική για αυτές τις διαπραγματεύσεις και σε σχέση με το ότι οι διατάξεις πνευματικής ε, ιδιοκτησίας ε, καλύπτουν, ωφελούν, διέπουν τους Ευρωπαίους πολίτες. Για την Νότια Κορέα, έχω να σας πω ότι υπάρχουν νόμοι εκεί που φιλτράρουν, που εμποδίζουν την επικοινωνία που παραβιάζουν τα δικαιώματα δημοτικής διευθυνσίας Αυτό δεν είναι καλό. Το ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν το μελετά, δεν το εξετάζει. Μια που στην υπόθεση Σαμπάμ έχει αποφανθεί σχετικά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Φυσικά και ο περιορισμός του, του ίντερνετ είναι φραγμός στην άσκηση εμπορία στο, στο, στο, όπου θέλει τελικά άρνηση του δικαιώματος του να ε, εμπορεύεται κανείς. 19 Ιουλίου είναι η προθεσμία της τροπολογίας και θα ψηφίσουμε στη συνεδρίαση της 17ης και 18ης Σεπτεμβρίου. Σας ευχαριστώ. 11. Δραστηριότητες ομάδων δραστηριότητες μάλλον υποπτικής ομάδα. Κίνα. Helmut Σόλτς. Να σας πω ποιο λόγια όσον αφορά την εποπτική ομάδα και την Κίνα. Χθε έγινε η τέταρτη συνάντηση με την εποπτική ομάδα. Ε, ασχοληθήκαμε με κάποια ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την τελευταία κοινή συνάντηση της 31ης Μαΐου εδώ στις Βρυξέλλες όπου παρέστηκε ο κύριος Ντεχίχτ και ο εμπορικός ακόλουθος της Κίνας Μας ενημέρωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτές τις ε, επαφές οι οποίες έγιναν με ειλικρίνεια, με πνεύμα ανοιχτό και οι δύο πλευρές ξέφασαν την υπεποίθησή τους ότι θα υπάρξει ευκαιρία να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία για τις επενδύσεις και θα γίνει αυτό φέτος το οποίο θα το φροντίσουμε Επίσης θα προχωρήσουμε παράλληλα με την ε, συνάντηση κορυφής 18-19 Σεπτεμβρίου, συνάντηση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Κίνας. Σύντομα δηλαδή. Και στα πλαίσια αυτής της συνάντησης θα αναφερθεί με προτεραιότητα ή εν λόγω συμφωνία. Επίσης, η ανταλλαγή απόψεων για τον νέο σύστημα άσκησης εμπορίας, συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ε, και αυτό αφορά Κίνα και Ιαπωνία. Αλλά έχει βεβαίως σημασία γενικότερα. Επίσης, Έχουμε και συμφωνίες Κίνας με Αυστραλία και Πακιστάν. Έχουμε επομένω μια στροφή της Κίνας που προσπαθεί επί τη βάση των συμφωνιών να ρυθμίσει τα θέματα συναλλάγματος και ισοτιμιών με αυτές τις χώρες. Απομένει να δούμε στο μέλλον ποιες θα είναι οι επιπτώσεις. Βεβαίως να δούμε και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομική κρίση. Πιστεύω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε στο τι θα γίνει με την εποπτική ομάδα. Οι συντονιστές να δούμε πώς θα συναρθρώσουν την προσπάθειά μας ε, εκεί. Σε σχέση λοιπόν με την δουλειά της ε, Επιτροπής Εμπορίου. Ο Πρόεδρος, συγγνώμη που δεν μπορούσα χτες να παραστώ. Τζόρτζ για το Μεξικό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους όσους όσοι χθε ήρθατε στην εποπτική ομάδα. Ήταν η πρώτη συνάντηση Επρόκειτο για πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση τον κύριο Γιώργεσεν και τον κύριο Ρωμάνγκο από την ε, Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Επρόκειτο για μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου πάρα πολύ φιλόδοξη. Αφορούσε όχι μόνο εμπορεύματα, αλλά και διευκόλυνση εμπορίου, τελωνιακά, δημόσιες συμβάσεις Έχουν κάποιο κύκλο ζωή βέβαια οι συμφωνίες αυτές. Επιδέχονται βελτιώσεις. Κολομβία, Νότια Αμερική έχουμε καλύτερε, πιο φιλόξε συμφωνίε. Έχουμε τρει ρήτρε αναθεώρηση που αφορούν για τη γεωργία, αφορούν τι επενδύσει. Πάντω θα ήθελε η Επιτροπή να αναθεωρήσει και επίση ε, και τις διατάξεις για τις δημόσιες συμβάσεις. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει συμφωνία σε σχέση με το πώς θα προχωρήσουμε προς αυτήν την αναθεώρηση. Η μεξικανική πλευρά δεν θέλει να εμπλακεί τόσο πολύ όσο εμείς, όσο θα ήθελε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντως, ε, θα πρέπει να μην ξεχνούμε ότι έχουν εκλογές, Τώρα θα ξεκινήσει ο διάλογος και έχουμε διάφορα άλλα θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί στην εποπτική ομάδα. Αυτά αφορούν την καταπολέμηση των ναρκωτικών, το ξέπλυμα του χρήματος. Όπως σας είπα, ήταν υπέροχη συζήτηση. Και Περιμένουμε ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις εξελίξεις στους αμέσως επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. We move on to Russia. Ρωσία. Έγινε η πρώτη συνάντηση με τον πρέσβη τέλος Ιουνίου και να πώς να το πω, να το διατυπώσω όσο μπορώ πιο προσεκτικά ήταν δύσκολο να του αποσπάσουμε μία απάντηση. Απέφυγε να απαντήσει στα περισσότερα. Αυτό ότι πάνε να πει βέβαια είναι καλός διπλωμάτης, ε? για τη χώρα του. Πάντως ένα από τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν ε, ε εκτενώς ήταν τα θέματα της κύρωσης της ε, αίτησης της Ρωσίας για τον ΠΟΕ. Βεβαίω και δεν υπάρχει ομοφωνία, αλλά το κόμμα του κυρίου Πούτιν θα κερδίσει και θα μπει στην Τούμα. Επίσης για το φυσικό αέριο. Δεν θα ολοκληρωθεί η κατασκευή του αγωγού και η γεωργία συζητήθηκε διότι Βεβαίω είναι τεράστιο εξαγωγέα η Ρωσία. Είχαμε μια-δυο κακέ οδιέ, αλλά θα συνεχίσουν ε, τι μαζικέ του εξαγωγέ. Ε, συζητήσαμε και τα θέματα θεώρηση διαβατηρίων. Βίζε για είσοδο στην Ρωσία. και έχει καταλήξει βέβαια μα είπε ότι πιο εύκολη είσοδο ε, στη Ρωσία από ό,τι στη ΣΥΠΑ είπε απάντησε σε ένα-δύο θέματα. Παρ' όλα αυτά. Τέλο πάντων, γενικά ε, είπαμε ότι ήταν πάρα πολύ ευχάριστη η συνεργασία. Και να δούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον. Δεν σχόλια. Καλώ. Επομένω, τώρα διακόπτουμε μέχρι τις 11.30. Έχουμε τους συντονιστές και κλεισμένων. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Και καλή όρεξη. Ποιος είναι ο Ρότζερ.